sì. Colleghe e colleghi, prendiamo posto. Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Πέρυσι, ξέρουμε τι έγινε στο Στρασβούργο όταν συνεδριάζαμε σε Ολομέλεια. Θυμούμαστε σήμερα λοιπόν τους νεκρούς των τρομοκρατικών και ισλαμιστικών αυτών επιθέσεων. Αντώνιο Μεγκαλίτσι. Ιταλός δημοσιογράφος που ήταν στο Στρασβούργο για να καλύψει την επικαιρότητα, την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και άλλοι από το Στρασβούργο, πολωνική υπηκότητα Γιαννιέ, Κανάλ Μπαγκάντ επίση, ε, δούλευε σε συνεργείο από το Στρασβούργο, αφγανικής καταγωγής. Πασκάλ Βερντέν επίσης, συνταξιούχος. Αμκουάνκ Σαμπέ Σαμάρνα, από την Ταϊλάνδη, τουρίστας στο Στρασβούργο. Η τρομοκρατία όμως δεν κοιτάει προέλευση. Κάνει μόνο θύματα και χτυπάει ολόκληρη την κοινωνία μας. Απέναντι λοιπόν στη βία και στον τρόμο, εμείς πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να στηρίξουμε τις ελευθερίες, τις αξίες που ουσιαστικά συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράζουμε λοιπόν την ελεγγύη μας, το σεβασμό μας σε όλα τα θύματα και στις οικογένειές τους, ε, τους φίλους του Στρασβούργου και ολόκληρο το γαλλικό λαό. Προτείνω λοιπόν ένα λεπτό σιγή προς τη μνήμη τους. Merci. Άρχονται λοιπόν οι εργασίες και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον, στην κυρία ε, Σινάτσοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ε, τσέχικα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από τις εργασίες ε, της ε, σημερινής συνόδου επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα τραγικά γεγονότα, στα θύματα ε, που υπήρξαν εχθές στην Τσεχία. Έξι σκοτώθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Οστράβα. Αυτό άνθρωποι που δεν θα επιστρέψουν ποτέ στι οικογένειές τους και στους φίλους τους. Είναι μια τραγωδία που δεν έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ. Ε, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στι οικογένειε του ε, και θα ήθελα επίση να σας παρακαλέσω να μεταφέρετε τα ε, συλληπιτήριά μα κι εσείς. Η κυρία Ελένα Λίτσι έχει το λόγο. Παρακαλώ. Καλημέρα Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου αφιερώνετε γιατί θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο έργο ενός ε, συμπατριώτη μου Ιταλού ο οποίος ήταν ο πατέρας του προγράμματος Εράσμους. Ήταν λοιπόν ένας αδελφός αν θέλετε αυτής της Ολομέλης. Ντομένικο Μαντούτσι πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία 86 ετών και φαντάζομαι θα ε, μπορείτε να φανταστείτε ότι αφήνει στην οικογένειά του ένα αναπλήρωτο κενό γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ δυνατός με διάθεση για πολλές πρωτοβουλίες αλλά αφήνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ε, ανεξίτηλη μνήμη για το τι μπορεί να είναι ένα πραγματικό κοινό εγχείρημα το οποίο μπορούν να μοιραστούν όλοι ακόμα ε, και το πώς μπορεί κανείς ε, να βλέπει στο μέλλον, μακριά στο μέλλον. Ίσως λοιπόν η Ολομέλειά μας ε, θα μπορούσε να τιμήσει τη μνήμη του και κάποια άλλη στιγμή στην Επιτροπή Απασχόλησης αυτό το ζήτησαν και άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να εκφράσω στην οικογένειά του, στις, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, τα συλληπιτήριά μας. Συμμετέχουμε στην, στο προσωπικό τους πένθος, αλλά θα ήθελα να έχω αναφερθεί εδώ σήμερα στον πατέρα του Εράσμους. Ήθελα να ε, τον έχω αναφέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάει λοιπόν η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, σταμάτησε στις 28 Νοεμβρίου. Ε, τα κείμενα της συνεδρίασης της 28 Οκτωβρίου. Τα πρακτικά υπάρχουν. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, αν δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε για τα πρακτικά, τα πρακτικά εγκρίνονται. Και κάποιες ανακοινώσεις μετά από την, ε, τον διορισμό της ε, κυρίας του Μπράσκα Σουίτσα, ε, της Αντίνα Ιωάννα Βάλεαν και του Νίκολα Σμιτ ως μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζει ότι χειρεύουν οι θέσει του από την 1η Δεκεμβρίου του 2019 και μονακίνωσαν οι αρμόδιε αρχέ την εκλογή των Σουκάνα Γκλάβακ που αντικαθιστά τον κύριο Σουίτσα και αναλαμβάνει ε, το αξίωμα από την 1η Δεκεμβρίου του 2019. Οι αρμόδιε υπηρεσίε τη Ρουμανία ενημέρωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον, ε, την εκλογή του κύριου Βλαντ Νίστορ ε, που αντικαθιστά την Αντίνα Βάλεαν από τις 2 Δεκεμβρίου του 2019. Οι αρμόδιες αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν την εκλογή του Μαρκ Άγγελ ε, στην θέση του Ευρωβουλευτή για αντικαθιστά τον κύριο Σμιτ από τις 10 Δεκεμβρίου του 2019. Βεβαίως ευχόμεθα σε όλους, ε, καλώς ορίσατε ε, και έχουν τα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς όλα αυτά που προβλέπει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη, τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Το τελικό σχέδιο καθορίστηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 28 Νοεμβρίου με βάση το άρθρο 157. Η ημερήσια διάταξη σας έχει διανεμηθεί. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, ε, επιθυμίε για τροποποίηση Η ομάδα των Πρασίνων συζήτησε η συζήτηση για τη δήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Συμφωνία να ολοκληρωθεί με ένα ψήφισμα που ε, θα τεθεί για ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λάμπερτ για να παρουσιάσει το αίτημα των Πρασίνων. Παρακαλώ, κύριε Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ζούμε μια πολύ σημαντική στιγμή. Είναι η πρώτη πολιτική πράξη της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει μεγάλη σημασία γιατί επηρεάζει όλες τις στι ευρωπαϊκές πολιτικές. Και χαίρομαι που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει και να παρουσιάσει σε εμά πρώτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την συμφωνία αυτή. Έτσι πρέπει να γίνεται σε μια κανονική δημοκρατία. Και πρέπει και εμεί να ανταποκριθούμε με ένα ουσιαστικό κείμενο, με ένα ψήφισμα δηλαδή στην πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να παρουσιάζει το όρομα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στι γενικέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εννοείται ότι θα έχουμε την ευκαιρία να αποφανθούμε για κάθε μία ε, χωριστά νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά είναι σημαντικό να δώσουμε και μια γενική άποψη ε, απέναντι σε ένα γενικό σχέδιο, μια γενική πρόταση που θα ακούσουμε. Και ελπίζω αυτό να γίνει, να εγκριθεί για την Ολομέλεια την 1η του Ιανουαρίου. Επιθυμεί κανεί ε, να λάβει το λόγο, διαφωνεί, ε, δεν υπάρχει κανείς να διαφωνεί. Ε, περνάμε λοιπόν στο αίτημα που ετέθη όποιος συμφωνεί ε, να σηκώσει το χέρι παρακαλώ όποιος συμφωνεί με τον κύριο Λάμπερτ κατά ε, όσοι διαφωνούν αποχές εγκρίνεται Άρα δηλαδή η συζήτηση για τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα επί το οποίο θα υπάρξει ψηφοφορία στην πρώτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορίστηκε λοιπόν η μερίσια διάταξη και περνάμε τώρα στην ε, ε, διακήρυξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Συμφωνία. Θα θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Φονταλάιν να την ευχαριστήσω καταρχήν για την παρουσία της εδώ και να της δώσω το το λόγο για να μας εισαγάγει στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδε έκανα μία υπόσχεση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας υποσχέθηκα ότι η Επιτροπή μου δεν θα χάσει χρόνο. Και να, δύο εβδομάδες ούτε καν αργότερα βρισκόμαστε εδώ ενώπιόν σας με την πρότασή μας για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, European Green Deal. Όντως, οι Ευρωπαίοι μας ζήτησαν να οδηγηθούμε σε μια αποφασιστική σημασία συμφωνία για το κλίμα. Και ακούγεται η φωνή των πολιτών και στους δρόμους αλλά και στις κάλπες. Και στο όνομα αυτών βρισκόμαστε εδώ σήμερα και στο όνομα αυτών παρουσιάζουμε αυτήν την πράσινη συμφωνία για την Ευρώπη που είναι τόσο φιλόδοξη. Σήμερα λοιπόν τους λέμε ότι ναι, σας ακούσαμε. Ναι, σας ακούσαμε να μιλάτε ξεκάθαρα και δυνατά και να ποια είναι η απάντησή μας. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, τον Ιούλιο, αμέσως αφού ορίστηκα σε αυτή τη θέση, έβαλα το σχέδιο για το κλίμα στο κέντρο της πολιτικής μας. Και εσείς με την δικιά σας ψήφο εγκρίνατε το πρόγραμμα αυτό. Σας υποσχέθηκα επίσης ότι εσείς θα είχατε μια κεντρική θέση στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Σήμερα ο Φρανς και εγώ και όλο το Σώμα των Επιτρόπων παρουσιάζουμε σε εσά αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες τις ιδέες μας για την Πράσινη Συμφωνία της Ευρώπης. Επίσης βρισκόμαστε εδώ επειδή σας χρειαζόμαστε. Η πρόταση αυτή δεν είναι το τελευταίο στάδιο της εργασίας, όχι, είναι η αρχή ενός κοινού δρόμου που θα διανύσουμε και αυτό μόνο μπορούμε να το κάνουμε με τη δικιά σας την υποστήριξη. Αξιότιμοι βουλευτέ. Δεν πρόκειται για ένα όραμα μόνο για μία ήπειρο ούτε τελείω που τον ε, κλίμα. Μιλάμε για ένα οδικό χάρτη με 50 πρακτικά βήματα για το δρόμο της Ευρώπης στο 2050. Θα μας πάρει πάνω από μία γενιά για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Το ξέρουμε ότι ο οδικό χάρτη αυτό θα πρέπει να εξελιχθεί και μάλιστα να προσαρμοστεί στην πορεία. Θα είναι μία μακρά διαδικασία και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν και εμπόδια. Αλλά σε εμά επαφείεται να θέσουμε το ρυθμό που θα ακολουθήσουμε και δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα πίσω. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι εφικτό είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε προς όφελος του πλανήτη και της ζωής στον πλανήτη αυτόν. Είναι τόσο πολλοί οι Ευρωπαίοι, οι πόλεις, οι επιχειρήσεις που μας καταδεικνύουν το δρόμο που θα ακολουθήσουμε την προηγούμενη Παρασκευή. 44 από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Ευρώπης που εκπροσωπούν 6-3 ευρώ σε ό,τι αφορά το αποθεματικό τους κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν ένα κλιματικό νομοθέτημα για τις προκλήσεις για το κλίμα μέχρι το 2050. Θέλουν να υπάρξει το νομικό αυτό πλαίσιο και λένε ότι θα τους δώσει την απαραίτητη εμπιστοσύνη για να λάβουν αποφάσεις μακροπρόθεσμες για τις σύγχρονες επενδύσεις. Είναι θέμα λογοδοσίας και αξιοπιστίας, ξέρετε και γι' αυτό αποτελεί ένα βασικό στοιχείο του, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα είναι το 2020 η πρόταση του πρώτου νομοσχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Θα θέσει σαφείς στόχους και ρόλους προκειμένου οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η μετάβαση επίσης προς την ουδετερότητα την θα είναι κάτι το αξιόπιστο. Και το επόμενο καλοκαίρι θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο για να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας για τη μείωση των εκπομπών. Αυτή η απόφαση για τους στόχους για το 2030 δεν θα είναι κάτι το τυχαίο. Το σχέδιο θα έχει μία πλήρη μελέτη αντικτύπου για να καταλάβουμε πού μπορούμε να είμαστε τολμηροί και πού πρέπει να είμαστε σόφρονες. Θέλουμε να είμαστε όσο φιλόδοξοι μπορούμε. Και θέλουμε να είμαστε και σωραλιστές γίνεται όλα αυτά θα είναι έτοιμα για την επόμενη COP26 στη Γλασκόβη. Η Ευρώπη θα ηγηθεί μέσω του παραδείγματός της, αλλά χρειαζόμαστε και πιο φιλόδοξου ε, πολυμερεί ε, κανόνες για όλο τον κόσμο. Φυσικά, κάθε ήπειρο θα πρέπει να βρει το δικό τη ε, δρόμο. Αυτό δεν χωράει αμφιβολία, αλλά ο στόχο θα πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους. Και η θετική αλλαγή θα πρέπει να ανταμείβεται, όχι να παρεμποδίζεται. Θέλουμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Καλωσορίζουμε την αλλαγή στην παραγωγή. Αν οι επιχειρήσεις επενδύουν στην πράσινη τεχνολογία, αν οι επιχειρήσεις σέβονται το περιβάλλον μας, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουν ε, ανταγωνισμό αυθέμητο από τους μεγάλους ρηπαντές και γι' αυτό λοιπόν έχουμε το μηχανισμό για την προσαρμογή των ε, στοιχείων αυτών ε, σε πλήρη συμβαδίζοντα πλήρω με τις ε, προδιαγραφέ του ΠΟΕ. Αξιότιμοι βουλευτέ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν αφορά μόνο τι εκπομπές. Έχει να κάνει με την ενίσχυση της ε, κοινοτομία, Έχει να κάνει με την ποιότητα. Έχει να κάνει με την σύγχρονη κινητικότητα. Και θα δημιουργήσει νέες αγορές και νέε επιχειρήσει σε όλη την Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα στρατηγική για την ανάπτυξη. Και η στρατηγική αυτή για την ανάπτυξη αυτή τη φορά δεν θα είναι κάτι που θα τα καταναλώνει μόνο, αλλά θα δίνει πιο πολλά από αυτά που παίρνει. Πρόκειται για μια στρατηγική για την ανάπτυξη η οποία θα έχει πιο πολλά στοιχεία όπως χρειάζονται. Οι επιχειρήσεις σε όλη την Ήπειρο στρέφονται προς την πράσινη μετάβαση, στρέφονται προς τις πράσινες ε, επιχειρηματικές ευκαιρίες. Κάποιοι ε, μετατρέπουν τα πλαστικά απορρίμματα σε σύγχρονα έπιπλα. Οι αγρότες χρησιμοποιούν δεδομένα από τους δορυφόρους για να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος μπαταρίες από την Ευρώπη για την ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα επιτέλους γίνονται πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στο δυναμικό της Ευρώπης για καινοτομία. Πριν από 70 χρόνια οι Ευρωπαίοι επένδυαν ε, στον χάλβα και στον ε, άνθρακα. Ήταν μια ιστορική συμφιλίωση και ένα οικονομικό θαύμα. Σήμερα επενδύουμε στις ανανεώσιμες ενέργειες και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει να κάνει ακριβώ με τη συμφιλίωση τη οικονομία μα με τον πλανήτη μα. Επανασυμφιλίωση λοιπόν με τον τρόπο που παράγουμε, με τον τρόπο που καταναλώνουμε στον πλανήτη μα. Και με το σεβασμό του περιβάλλοντο στο οποίο ζούμε. Αυτό είναι ο πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αξιότιμοι βουλευτέ. Πριν από ένα ακριβώ χρόνο, η πόλη του Κατοβίτσε υποδέχτηκε το παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα, COP24. Η πόλη λοιπόν αυτή, η οποία για πάνω από ένα αιώνα ήταν η πρωτεύουσα του άνθρακα, έγινε η παγκόσμια πρωτεύουσα της κλιματικής δράσης. Αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο από τις πρώινα βιομηχανίες του άνθρακα που πλέον έχουν συνέδρια, εστιατόρια, μέγαρα αυτή η μετάβαση δεν έγινε σε μία νύχτα. Και δεν έγινε χωρίς κόπο. Παρομοίω, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν πρόκειται ούτε αυτή να πραγματοποιηθεί σε μία νύχτα και θα είναι πολύ απαιτητική. Αλλά είναι ο σωστό δρόμο. Όπω και στο Κατοβίτσε, η μετάβαση θα επιφέρει πιο καλέ, πιο υγιεί θέσει απασχόληση, πράσινε, ε, λιγότερο βρώμικες πόλεις, για ποιότητα ζωής για όλους τους Ευρωπαίους. Αυτή η μετάβαση όμως θα πάρει χρόνο. Υποστήριξη και αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν του χρόνου κατευθείαν θα προτείνουμε το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης που θα συνδυάζει δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρησιμοποιηθεί ως μόχλαυση για να πετύχουμε τα 100 δις ευρώ σε επενδύσεις τα επόμενα 7 έτη. Θα αποτελέσει λοιπόν το εφαλτήριο για τις ε, επιχειρήσεις αυτές και τις ε, περιοχές που θα πρέπει να επιταχύνουν. Όλοι στην Ευρώπη λοιπόν μπορούν να είναι τμήμα της αλλαγής αυτής. Η μετάβαση αυτή δεν αφορά μόνο ε, τις μεγάλες βιομηχανίες και τον άνθρακα. Αποτελεί μια ευκαιρία για τους αγρότες μας σε ό,τι αφορά τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο, από τη Λαπωνία μέχρι την Νότια Ιταλία. Μια ολόκληρη γενιά νέων αγροτών ανακαλύπτουν εκ νέου παραδοσιακούς τρόπους και παραδοσιακά είδη. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Πράσινη Συμφωνία θα είναι στο πλευρό τους και θα φροντίσει τους απίστευτους ε, φυσικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προωθήσει την βιοπικιλότητα και θα προωθήσει και την πράσινη οικονομία. Εμείς όμως ως θεσμικά όργανα που είμαστε στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Και αυτό θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει επίσης να μάθουμε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή στην καθημερινή μας ζωή. Πώς μπορούμε να είμαστε πραγματικά βιώσιμοι. Τι σημαίνει να έχουμε τα σωστά κτίρια για τα απορρίμματά μας, για τα ταξίδια μας, για τη χρήση χαρτιού, για όλα. Σήμερα λοιπόν στο Σώμα των Επιτρόπων θέτουμε το στόχο ως Επιτροπή να είμαστε μέχρι το 2030 κλιματικά ουδέτεροι και καλό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να κάνουν το ίδιο. Είναι πρόκληση, αλλά ας την αντιμετωπίσουμε μαζί. Να υποστηρίξουμε λοιπόν τους ενεργούς πολίτες και να ζητήσουμε να προωθηθούν αυτές οι πρωτοβουλίες τους, να συνεργαστούμε με τους δασκάλου, ε, του ε, δασκάλους, τους καθηγητές, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι παθητικοί παρατηρητές, είναι πολύ ενεργοί φορείς σε αυτή τη διαδικασία. Το πράσινο αυτό σύμφωνο, η πράσινη συμφωνία θα είναι μια συμφωνία μαζί τους και για αυτούς, για όλους όσους είναι έτοιμοι να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, αξιότιμοι βουλευτές όλη η Ήπειρος θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Από τους δημάρχους στις μικρές πόλεις και στις μεγάλες πόλεις σε, μέχρι όλα τα θεσμικά όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα τα μέλη της Επιτροπής μου θα συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή, όλα τα κράτη-μέλη, κάθε επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο. Και μάλιστα όλα αυτά δεν μπορούν να είναι δυνατά χωρίς την υποστήριξή σας. Θα χρειαστούμε φιλόδοξη νομοθεσία θα, χρειαστούμε έναν επτάτη προπολογισμό ο οποίο θα ταπεξέλθει στον ύψο των προκλήσεων. Σήμερα λοιπόν φέρνουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Αύριο θα την παρουσιάσουμε στους ηγέτες στο Συμβούλιο. Και αργότερα, μέσα στην εβδομάδα, ο Φραντ Τίμερμαν θα τα παρουσιάσει αυτά στην Μαδρίτη στο COP25. Α ξεκινήσουμε λοιπόν από κοινού αυτό το εγχείρημα. Αξιότιμοι βουλευτέ. Κάποιοι διατείνονται ότι το κόστος της ε, μετάβασης αυτής, της μεταμόρφωσης αυτής είναι πολύ υψηλό. Ας μην ξεχνούμε όμως ποιο είναι το κόστος της μη ανάληψης δράσης. Αυξάνεται κάθε χρόνο οι πλημμύρε ε, κοστίζουν κάθε χρόνο πάνω από 5 δισεκατομμύρια και κάθε χρόνο η οικονομία μας χάνει περίπου 10 δις ευρώ λόγω της ξηρασίας και το πιο υψηλό τιμήμα το πληρώνουν οι αγρότες. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο. Μπορούμε να αντισταθούμε στις εξελίξεις αυτές έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, αλλά δεν είναι πολύ αργά. Με τον οδικό χάρτη αυτό για τη δράση κάνουμε το κόστος της πράσινης μετάβασης βιώσιμο και πολλοί Ευρωπαίοι ήδη αναλαμβάνουν δράση. Πριν από ένα έτος μόλις, κανείς δεν θα φανταζόταν ότι εκατομμύρια θα βγαίνουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν υπέρ του περιβάλλοντος. Οι πολίτες μας επιλέγουν την καθαρή ενέργεια, οι επιστήμονες αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του μέλλοντος, οι οικογένειά μας σταματούν να χρησιμοποιούν το πλαστικό και επιλέγουν τα τοπικά προϊόντα και τρόφιμα. Αυτή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία λοιπόν είναι για αυτού. Είναι φιλόδοξη. Έχει σχεδιαστεί με δίκαιο τρόπο. Είναι made in Europe. Φτιαχμένη στην Ευρώπη για την Ευρώπη για να μα οδηγήσει μέχρι την κλιματική ιδιωτερότητα μέχρι το 2050. Η Ευρώπη πάντα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε σε... όταν εργαζόταν από κοινού ως Ένωση. Εμείς λειτουργούμε καλύτερα όταν είμαστε τολμηροί και έχουμε υψηλούς στόχους. Και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτουμε υψηλούς στόχους. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν μας ζητούν να είμαστε εμείς η κινητήρια δύναμη της αλλαγής αυτής. Τώρα από εμά επαφείτε να πραγματοποιήσουμε αυτή την αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Και τώρα λοιπόν ε, θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ε, κυρία Ντελάγκε. Παρακαλώ, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που σήμερα μας παρουσιάσετε το όραμα, τα προγράμματα και τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία. Για το ΕΛΚΑ, για μας, για τα λαϊκά κόμματα, τους Christian Δημοκράτες, τα κίνητρά μας είναι απόλυτα σαφή. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μας ανήκει ο πλανήτης, απλά τον φροντίζουμε για την επόμενη γενιά. Και έχουμε και την ηθική υποχρέωση να τον προστατεύσουμε. Άρα δηλαδή Αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα για μας δεν είναι απλά μια συμφωνία, είναι μια ε, υπόσχεση προς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αναφέρθηκε ε, στο ότι επιδιώκουμε κάτι ε, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό απαιτεί βεβαίως τάρος αλλά σημαίνει και ότι πρέπει να δράσουμε. Ίσως να είμαστε η τελευταία γενιά που να μπορεί να δραστηριοποιηθεί και αυτό να κάνει κάποια διαφορά. Ε, έχουμε κάποιες δεκαετίες μπροστά μας που πρέπει να επιτύχουμε στόχους. Βεβαίως, αναφέρθηκε η ότι δεν μπορούμε να στείλουμε ανθρώπους στο διάστημα με το να θέλουμε θέλουμε να επιβάλλουμε στους άλλους το τι δεν πρέπει να κάνουν. Αυτό που θέλουμε είναι να ενώσουμε τους καλύτερους, τους πιο ευφυείς. Χρειαζόμαστε ρήξη και έλευτες λύσεις, την καθαρή βιομηχανία που θα προσφέρει θέσεις απασχόλησης στους νέους και ευκαιρίες. Η Ευρώπη λοιπόν ας είναι ήπειρος εκείνη η οποία θα παράγει εναλλακτικά κάψιμα για τα αεροσκάφη και να περιορίζει και τις διαδρομές. Ας είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα παράγουν ε, λιγότερο χάλιβα. Ίσως ε, εμείς στο ΕΛΚ να μην είμαστε πολεμιστές ε, για το κλίμα, αλλά είμαστε εκείνοι που πραγματικά νοιαζόμαστε. Και αυτό χρειάζεται η Ευρώπη. Το δεύτερο που θα κάνουμε είναι να μην θέλουμε να μείνει κανείς παραμελημένος. Παραδείγματο χάρη, δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε εκείνου που δεν είναι σε θέση να φέρουν το βάρος. Και αυτό πραγματικά ανησυχεί τους Ευρωπαίους. Αυτό το κάνουμε συνεργαζόμενοι με, τους, με τα, ασχολούνται με τα δάση, με τους αγρούς, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι εκτάσεις αυτές στην Ευρώπη και αυτό είναι πραγματικά ε, ένα ε, κομμάτι του προβλήματος. Εκεί είναι και η λύση να τους προσφέρουμε καλές τιμές για τα προϊόντα τους ε, και, ένα, και πολύ καλούς ίσως όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Επίσης να είμαστε συνεπείς. Για το ΕΛΚ είναι απόλυτα σαφέ ότι μια φιλόδοξη πολιτική κλίματος και μια ευφυή σε βιομηχανική πολιτική πρέπει να συμβαδίζουν. Πράσινη συμφωνία χωρίς καλή συμφωνία για τη βιομηχανία μας δεν θα επιφέρει την αλλαγή που αναζητάμε. Θέλουμε λοιπόν και χρειαζόμαστε φιλοδοξίες ε, και ένα επιχειρηματικό πλαίσιο ε, και ίσως όρους ανταγωνισμού. Αναφέρθηκε ότι άλλα μέρη του κόσμου ε, δεν μπορούν να έχουν κάποια πρόσβαση, διορθωτική πρόσβαση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Σήμερα νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την κατεύθυνση που ακολουθούμε. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, αλλά η δουλειά του πώ θα φτάσουμε εκεί τώρα ξεκινάει. α μην αυταπατώμεθα, δύσκολα όλα αυτά. Χρειαζόμαστε συνδυασμό οράματο και πρακτική στρατηγική. Και ακριβώ αυτό μπορεί και θα κάνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η πρόεδρος Γκαρσία Πέρες, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και εσεί, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή για την Ευρώπη και για τον πλανήτη μα. Λίγε μέρε μόνο μετά από την έναξη εντολή επιτροπή, χάρη στην εξαιρετική εργασία του φραντ Τίμερ μα, μα παρουσιάζει σήμερα κάτι παραπάνω από μια πρόταση. Σήμερα μα παρουσιάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξη που έχει όσο στόχο να τροποποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την καταστήσει μια πιο δίκαια κοινωνία, περισσότερο ευημορούσα που θα μπορέσει να απαντήσει στι προκλήσει Τη της κλιματικής αλλαγής. Τον Νοέμβριο που μας πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι επήγει η υπόθεση του κλίματος. Για τους σοσιαλδημοκράτε δεν πρόκειται για ένα κενό περιεχομένου σλόγγαν. Πρόκειται για μια προειδοποίηση που απαιτεί επιγόντω μέτρα και έκτακτα μέτρα. Η Πράσινη Συμφωνία λοιπόν δείχνει το δρόμο που πρέπει να διανύσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπο κόσμο για να υπάρξει μετάβαση αυτή. Αποτελεί ένα πρότυπο για να μπορέσουμε επιτέλου να σταματήσουμε με τα στερεά ορυκτά και να έχουμε μια Ευρώπη που θα είναι ουδέτερη όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα το 2050. Χρειάζεται όμω μια δίκαια μετάβαση με τρει πυλώνε. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα πράσινο πυλώνα που να εφαρμόζει του στόχου του 2030 30 των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα θεωρούμε πολύ θετική την ε, πρόταση επειδή ε, δίνει σάρκα και οστά τους στόχους μας που θέλουμε να συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και αναφέρομαι στον πράσινο πυλώνα για τη βάση συγκεκριμένου στόχου για το κλίμα και την δέσμευση να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Δεύτερο πυλώνα είναι ο κόκκινο πυλώνα, η κοινωνική διάσταση δηλαδή τη πράσινη συμφωνία. Στην Πράσινη Συμφωνία χρειαζόμαστε μια πραγματική κοινωνική διάσταση και αυτή θα την πετύχουμε με έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνα που θα μας επιτρέψει να τροποποιήσουμε τις οικονομίες μας και θα διασφαλίσει κανείς να μην μείνει ξεχασμένος πίσω. Δεν είναι δυνατόν ε, οι πιο αδύναμοι να πληγούν περισσότερο. Και ο τρίτο πυλώνας είναι ο οικονομικό που θα καθορίσει την επιτυχία τη πράσινη συμφωνία. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η υλοποίηση των στόχων χρειάζεται επιπλέον 260 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να πετύχουμε την συμφωνία αυτή. Χρειαζόμαστε 1,3% του ΑΕΠ και χρειαζόμαστε και δίκαια φορολογία επίσης που να ευθυγραμμίζεται με του στόχου μείωση χρήση του άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή μόνη τη όμως η εμπορική μα πολιτική ε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προωθήσουμε τι δικέ μα προδιαγραφέ, τι εργασιακέ, τι κοινωνικέ και τι περιβαλλοντικέ. Σήμερα λοιπόν στέλνουμε ένα σαφέ μήνυμα για να τηρήσουμε και να δώσουμε συνέχεια ε, στα όσα επιθυμεί ο κόσμο, ο οποίο βγαίνει στου δρόμου να διαδηλώσει υπέρ του κλίματο. Είναι έτοιμο ο κόσμο για τι αλλαγέ. Εμεί οι σοσιαλδημοκράτε επίση είμαστε έτοιμοι για την αλλαγή. Το ερώτημα είναι το εξή. Οι ηγέτε μα και οι υπόλοιπε πολιτικέ δύναμε είναι έτοιμε για την αλλαγή αυτή. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από το ναι είμαστε. Εκ μέρου τη ομάδα, Renew Europe, ο πρόεδρο κ. Ατσόλο. παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, η Πράσινη Συμφωνία είναι η αρχή μιας διαδρομής για να βρεθεί η Ευρώπη στο σωστό δρόμο να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Αλλά θα τα καταφέρουμε μόνο αν αυτήν την πρόκληση τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία για τους πολίτες και την οικονομία μας. Αν ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, η Renew Europe θα είναι αξιόπιστος αλλά και απαιτητικός εταίρος. Διαβάσαμε την διακήρυξη για την έκτακτη κλιματική ανάγκη ε, και θεωρούμε ότι η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να βρίσκεται σε πρώτη θέση στην ημερησία διάταξή μας. Πρέπει να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία. Η Πράσινη Συμφωνία δεν μπορεί να καταλήξει με περισσότερη γραφειοκρατία, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη κοινωνική δυναμική. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, αλλά και πρέπει να εμπλακούμε σε μια ευρύτερη συζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη για αυτό το εγχείρημα. Για να προκαλέσουμε αλλαγή, πρέπει οι φιλοδοξίε μα να ενταχθούν σε μελλοντική κλιματική νομοθεσία και να είναι ε, πάντα απαραίτητο να υπάρχει μελέτη αντικτύπων. Η μετάβαση προς την οικονομία ουδέτερη προς ε, εκπομπές, αυτό είναι μια ευκαιρία, βεβαίως απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, δημιουργικότητα, αλληλεγγύη με τους ανθρώπους και με τον τομέα που θα αντιμετωπίσουν την πιο δύσκολη μετάβαση. Το τρίτο, μια διτή προσέγγιση στην πράσινη ψηφιοποίηση και την τεχνολογία, αυτά είναι καθοριστική σημασία για μα. Οι ψηφιακέ τεχνολογίε είναι σε μοναδική θέση να προσφέρουν αποτελεσματικά εργαλεία για την άμπλυνση ε, και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και τέλο, η τέταρτο, δεν πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε, ε, σε νέε πολιτικέ. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε τι παραδοσιακέ μα, γιατί η κοινή γεωργική πολιτική μπορεί να συμβάλλει στου νέου στόχου. Οι νέε πράσινε φιλοδοξίε πρέπει να ολοκληρώνονται με πολιτικέ μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν προταθεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι η πρόκληση μιας ολόκληρης γενιάς, αλλά το ταξίδι μας μπορεί να είναι και ευκαιρία για την επανανακάλυψή μας. Ε, το δύσκολο δεν είναι μόνο να βάζει κανείς φιλοδοξίες, αλλά και να βρίσκει και πρακτικές λύσεις. Μπορείτε λοιπόν να μας εμπιστευτείτε. Εμείς ως Renew Europe θα είμαστε ένας πραγματικά δραστήριος εταίρος. Ο πρόεδρος κύριος Λαμπέρτς εκ μέρους των Πρασίνων. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καθιστά το οικολογικό ζήτημα ένα μεγάλο έργο το οποίο αναλαμβάνει. Και αυτό ακριβώ είναι η σημερινή Πράσινη Συμφωνία. Δέκα μέρε χρειάστηκαν για να προχωρήσει στο σχέδιο Επιτροπή. Το ερώτημα είναι τώρα να δούμε κατά πόσο και πώ αυτό ο κατάλογο καλών προθέσεων θα υλοποιηθεί και θα γίνει συγκεκριμένα έργα. Εμεί τέσσερα κριτήρια βλέπουμε για την Πράσινη Συμφωνία. Πρώτον, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά αγωνίζεται για να καταπολεμήσει την ε, θέρμανση του πλανήτη για να περιοριστεί κάτω από τον 1,5 βαθμό. Προ το παρόν πολλά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Τις επόμενες 100 μέρες λοιπόν πρέπει να δεσμευτούμε να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά 55% μέχρι το 2030. Η κλιματική απορρίθμιση αποτελεί μόνο ένα σύμπτωμα ε, του γεγονότο ότι η ανθρωπότητα δεν σέβεται τα όρια του πλανήτη. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε για την βιοπικιλότητα, για την εξάντληση των πόρων ή ακόμα και για την ε, ρήπανση τη φύση από την οποία εξαρτάται η ίδια μας η ζωή. Δεύτερον, για να πετύχουμε την ε, οικολογική μετάβαση πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Πρέπει συγχρόνως να μειωθούν οι οικονομικές και οι κοινωνικές ανισότητες. Εννοείται ότι το να παράγουμε και να καταναλώνουμε με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον κοστίζει πιο ακριβά. Το να τα βάλουμε όμως ε, τον φόρτο σε αυτούς που υποφέρουν από τη φτώχεια δεν είναι δίκαιο και μας το έχουν υπενθυμίσει αυτό τα κίτρινα γυλαίκα. Επίσης, αν ε, θέλουμε, μάλλον εφόσον πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει και θέσει απασχόληση η μετάβαση αυτή, να ξέρουμε ότι θα καταστρέψει κιόλα. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα και γι' αυτό χρειάζεται αλληλεγγύη και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να επιβραβεύουμε αυτούς που χρησιμοποιούν τα αστερά κάψιμα, αντίθετα. Και χρειάζεται μια δίκαιη απάντηση, χρειάζεται μια μετάβαση σε βάθος και της φορολογίας, ώστε όσοι έχουν υποφεληθεί από τα αστερά κάψιμα μέχρι τώρα να είναι αυτοί που θα πληρώσουν και το τίμημα της μετάφασης. Τρίτον, η Πράσινη Συμφωνία απαιτεί συνέπεια από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, γιατί τι νόημα έχει να δίνουμε ένα τέταρτο του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσουμε την κλιματική απορρίθμιση, αν τα υπόλοιπα τρία ε, τέταρτα ε, πηγαίνουν σε δράσει οι οποίε ακριβώ επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε με μια πολιτική η οποία βασίζεται στην παραγωγικότητα και όλο και περισσότερη παραγωγικότητα υπέρ των ε, παγκοσμίων αγορών. Και τι να πούμε και για τι ελεύθερε συναλλαγέ στην Ένωση. Το να αυξάνονται όλο και περισσότερο οι εμπορικέ συναλλαγέ είναι κάτι που καταστρέφει το περιβάλλον. Οπότε ε, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δούμε τις ε, αντιφάσεις, κάτι που προσπαθείτε να κάνετε, αλλά πρέπει να είμαστε και πιο αποφασισμένοι. Τέλος, δεν έχει πιθανότητες επιτυχίες η Πράσινη Συμφωνία αν δεν βάλουμε την οικονομία ε, στην υπηρεσία της κοινωνίας. Γιατί από το 2007 πρέπει να ξέρουμε ότι το DNA του θηρίου που είναι ο χωπαστοτικός τομέας και ευθύνεται για τα κακά που θέλει να καταπολεμήσει η Πράσινη Συμφωνία παραμένει ανελίωτο και αυτό είναι ανεύθυνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και 60 χρόνια για πρώτη φορά επιστήμονε άρχισαν να κάνουν τη σύνδεση ανάμεσα στι ανθρώπινε δραστηριότητε και την κλιματική απορρίθμιση. Και πριν από ε, πέντε χρόνια ο όμιλο τη Ρώμη μα έκλουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το θανάσιμο κίνδυνο τη οικονομική μεγέθυνση χωρί τέλο. Πριν από 30 χρόνια, στο Ρίο, ο Ζακ Σιράκ κατήγγειλε πω το σπίτι μα καίγεται και ότι εμεί πέρα βρέχει. 20 χρόνια μετά την πρώτη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, και οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους. Συγχρόνως εξαντλούνται οι πόροι μας και καταστρέφεται η βιοπικιλότητα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ετοιμαστούμε για τη μάχη. Γιατί αν, κυρία Πρόεδρε, γενικεύσουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη αυτό τον τρόπο ευρωπαϊκή ζωή που θέλετε εσεί να προωθήσετε, τότε ε, θα χρειαζόμασταν τέσσερι πλανήτε. Όχι έναν, έχουμε όμω έναν μόνο και από αυτόν εξαρτάται η ζωή μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, η κυρία Σερντόνε εκ μέρου τη ομάδα ID. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εκτό από το γεγονό ότι εγώ είμαι καινούργια εδώ, ε, ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ε, θα έπαιρνα τα έγγραφα στην αίθουσα και να ξέρω να συζητάω για αυτά. Σω ίσως ε, θα μπορούσε ε, κανείς να μας θα δώσει νωρίτερα για να διαβάσουμε κάτι. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η δημοκρατία σε αυτή την αίθουσα. Είναι πολύ δύσκολο να διαβάσει κανείς τα έγγραφα εκ των προτέρων έγγραφα για τα οποία καλύτερα να συζητήσει. Ε, μέχρι το 2050 υπάρχουν πάρα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. Η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 έτσι λέτε. Αλλά έχετε σκεφτεί τις επιπτώσεις τις κοινωνικές και τις οικονομικές. Κατανοώ βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θέλει να εμφανίστε κάπως μοντέρνα, αλλά δεν νομίζω ότι με το να βγάζει και να πετάει κανείς σλόγγαν ότι αυτός, αυτό είναι ο σωστός τρόπος. Έγινε λόγος ε, για την προαγωγή της ε, καινοτομίας ε, και της ποιότητας των τροφίμων. Αυτή η ποιότητα των τροφίμων είναι αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες, τα αφρικανικά ας πούμε πορτοκάλια. Στην Ευρώπη ζητάτε πρότυπα. Από την άλλη όμω βλέπουμε κατά κάποιον περίεργο τρόπο να συνάπτονται εμπορικέ συμφωνίε, ακόμα και με χώρε που δεν εφαρμόζουν αυτά τα πρότυπα. Ε, εκεί για τα πλαστικά συζητάτε χωρί πλαστικέ ουσίε και τι κάνετε, συνάπτεται εμπορικέ συμφωνίε με χώρε όπου η ρήπανση είναι στην ημερήσια διάταξη. Άκουσα ότι έγινε λόγο για μπαταρίε που κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα το 60% όλων των μπαταριών του κόσμου κατασκευάζονται στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα. Και άκουσα επίση ότι έχει υπάρξει πλέον μια εξέλιξη από τον άνθρακα στο χάλιβα ε, και τώρα είμαστε στην φιλοδοξία της παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο και διαρωτώ με ποια είναι η χώρα εκείνη η οποία τυχαία ίσω θα ήθελε να μετατρέψει το παραγωγικό σύστημα ει βάρο όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν ξέρω, ίσω αυτό να το υποψιαζόμαστε μόνο εμεί, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα μιλάνε από μόνα του. Μιλάτε για 100 δις επενδύσεις τα επόμενα 7 χρόνια και τελικά είσαστε εσείς οι ίδιοι οι οποίοι ψάχνετε ε, να βρείτε και το τελευταίο κόμμα στον προπολογισμό και αυτό σε σχέση με χώρες ε, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους ε, στον τομέα των υδάτινων πόρων. Και κάτι τελευταίο. Έχω την εντύπωση ότι για δεύτερη φορά άκουσα το πρόγραμμα Juncker, δηλαδή που μας είχαν τότε μιλήσει για τους πολλαπλασιαστές, ότι αν βάζαμε ένα ευρώ θα κερδίζαμε 1500 ε, περισσότερα. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Εύχομαι λοιπόν ότι να έχετε τη δυνατότητα να έχετε ένα ρεαλιστικό όραμα και να ξεφύγετε από τα συνθήματα τα οποία ε, παπαγαλίζεται ο σαν να ήταν καραμέλες. Από το ECR, ε, Λεγκούτκο παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τρία στοιχεία. Καταρχάς, πρώτο, συναντιόμαστε υπό έκτακτες συνθήκες. Συζητάμε τις αλλαγές που γίνονται στο κλίμα και στους ενεργειακούς στόχους αλλά δέκα ημέρες ε, μετά την ανάληψη των καθήκοντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν την εφαρμογή των υφιστάμενων ε, συμφωνιών για το κλίμα. Αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά δεν είναι σόφρον. Δεύτερο στοιχείο. Στο ECR ελπίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν λίγο πιο προσεκτική από την προηγούμενη. Ότι θα συνεργάζονταν με τα κράτη-μέλη και με τις ε, πόλεις και στο πλαίσιο των συνθήκων το άρθρο 15 αναφέρει με σαφήνεια ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό που ορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συναντηθεί αύριο για να συζητήσει τι την μακροπρόθεσμη πολιτική για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερωτώμε λοιπόν γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αφαιρέσει την ε, δύναμη και την εξουσία αυτή των κρατών μελών. Κοιτώντα αναδρομικά, είδαμε, βλέπουμε ότι το 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε. Οι στόχοι του 2030 να επιτευχθούν με συμβιβασμό μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και επίπονες και σήμερα μιλάμε για κλιματική ιδιωτερότητα μέχρι το 2050 θα έπρεπε να έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, την ίδια οδό και τα, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεν θα έπρεπε να παραγωνίζονται για κάτι τόσο βασικό. Τρίτο σημείο, κυρία Πρόεδρε. Πρόσφατα έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το πράσινο κύμα αυτό το οποίο περνάει την Ευρώπη. Αλλά προσέχετε μήπως ότι κάθε φορά που φτάνει στην Βαλτική και πάει στο Δούναβη δεν είναι καν ε, μικρό κύμα. Γιατί? Γιατί βλέπουμε μια στρατηγική που προκαλεί πιο πολύ σύγχυση και ερωτήματα παρά απαντήσεις. Οι νέοι στόχοι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιτεύξιμοι, είναι αξιόπιστοι. Τι θα κάνουν στις ε, βιομηχανίες μας. Μας δώσατε μια εικόνα ενός παραδείσου, μα ποιος δεν θα ήθελε να ζει στον παράδεισο. Αλλά πώς θα πείσει αυτό τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων η νέα επιτροπή σε δέκα μέρες από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά τη είναι σε θέση να κατανοήσει σε βάθος τη δραματική κατάσταση την οποία μπορούσε να επιφέρει αυτή η πράσινη συμφωνία στην οικονομία μας. Έχετε καθόλου ιδέα για το κοινωνικό κόστος, τι προσωπικέ τραγωδίε που θα συνεπαγόταν αυτό. Τέταρτο σημείο, το οποίο σκόπευα να το παραλείψω, αλλά θα το αναφέρω εν συντομία. Σε ό,τι αφορά το αέριο. Βλέπουμε εδώ μια πολύ περίπλοκη στρατηγική, γιατί το αέριο θα αποτελέσει βασικό τμήμα της μείωσης του ανθρακά και θα απαγορευτούν οι μελλοντικέ επενδύσεις από την άλλη αναφέρεται στο αέριο. Αυτό προκαλεί σύγχυση. Για να συνοψίσω λοιπόν κυρία Πρόεδρε. Το πώς θα κινηθούμε προς το, μπροστά θα πρέπει να προκαθοριστεί με αξιόπιστο τρόπο Ιδάλλως μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, να θέσουμε όποιο στόχο θέλουμε, δεν θα έχει καμία αξία αν δεν μπορούμε να τους πετύχουμε. Και αν προσπαθήσουμε να το επιβάλλουμε με τη βία, οι συνέπειες θα είναι ενδεχομένως καταστροφικές. Ευχαριστούμε ε, κυρία Ομπρί, εκ μέρους της ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση δεν είναι μια συνηθισμένη συζήτηση. Μιλάμε για κάτι πολύ σημαντικό που ξεπερνάει τις διακρίσεις μεταξύ μας και τις διαφορές. Έχει να κάνει με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη όπως τη γνωρίζουμε. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρόμαστε που ήρθε να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα δράσης της. Αλλά λέμε ευθύ εξ αρχής, κάθε κλιματική πρωτοβουλία θα είναι μάταιη αν δεν αντιμετωπίσει και τη ρίζα του προβλήματος ένα οικονομικό σύστημα το οποίο οδηγεί στην καταστροφή του οικοσυστήματός μας και σε αύξηση των ανισοτήτων. Κάποιες από τις προτάσεις σας όπως για την ανδάσωση, για τις κρατικές ενισχύσεις ή την ε, ενεργειακή μετάβαση κτλ. Είναι θετικά στοιχεία. Αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπουμε πώς θα χρηματοδοτηθούν και δεν είναι και υποχρεωτικά. Βλέπουμε πολλά προγράμματα, πολλά σχέδια δράση, στρατηγικέ που ανακοινώνονται, αλλά δεν βλέπουμε πραγματικέ νομοθετικέ αλλαγέ. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι με λόγια που θα σώσουμε το πλανήτη. Έπειτα υπάρχουν και αντιφάσει στι προτάσει σα με αποτέλεσμα κάποιοι στόχοι να μην μπορούν να υλοποιηθούν. Πώς είναι δυνατόν για την ενέργεια να μην έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή και πόσο περιμένουμε ότι θα πάψουμε να χρησιμοποιούμε τα αστεριάνθρακα άμα δεν ξέρουμε πότε. Αν συνεχίσουμε τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που οδηγούν σε τόσα προβλήματα, πώς είναι δυνατόν να μην ανοίγουν οι διαπραγματεύσει για νέα κοινή γεωργική πολιτική. Πώς είναι δυνατόν να καταστρέφουμε τις δημόσιες ε, επιχειρήσεις και να λέμε ότι θέλουμε περισσότερα τρένα. Πώς είναι δυνατόν να μην προτείνετε φόρο για τα πλαστικά, την τα κτλ. Και συνολικά δεν θα πετύχει ο στόχος σας για το 50% ε, μείωση των εκπομπών που προτείνεται που απαιτεί και Συμφωνία των Παρισίων. Και έπειτα κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη δικιά μας την ομάδα. Ξεχνάτε την ανθρώπινη και την κοινωνική διάσταση ε, της ε, οικολογικής μετάβασης, ενώ η ίδια παραδέχεστε ότι οι περισσότερο φτωχοί είναι και αυτοί που βρίσκονται σε περισσότερο επισφαλή θέση. Χρειάζεται ε, μια πολύ ισχυρή πολιτική απόφαση. Δεν θα αλλάξουμε την κλιματική κατάσταση αν το κάνουμε σε βάρος των ανθρώπων ή όπως προσπαθεί να το κάνει ο Μανουέλ Μακρόν στη Γαλλία. Η οικολογική μετάβαση πρέπει να γίνει από τον κόσμο και με τον κόσμο. Οπότε, ε, ότι επήγει, ναι, επήγει, αλλά χρειάζεται μια πραγματική νέα συμφωνία και κοινωνική και οικολογική η Ευρώπη. Ε, τεράστιων διαστάσεων που δεν είχαμε δει ποτέ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξού και η πρόταση τη ομάδα μου, τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, που σα υποβάλλουμε σήμερα και που καταθέτουμε με συγκεκριμένες προτάσεις που διαρθρώνονται γύρω από 10 άξονες. Πρώτα απ' όλα η Νέα Πράσινη Συμφωνία πρέπει να έχει ένα κλιματικό νόμο με στόχο και προτεραιότητες. Δεσμευτικό μείωση των εκπομπών 60% μέχρι το 2030 και επίσης με ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο ώστε να περάσουμε στο 100% ανανόσιμες πηγές ενέργειας το 2050 και με δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά την οικονομία ενέργειας από τις επιχειρήσεις. Επίσης πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα θερμικής ανανέωσης και ενεργειακής ανανέωσης ώστε να πάψουν να βρίσκονται στην ενεργειακή φτώχεια τα εκατομμύρια των συμπολιτών μας. Πρέπει να υπάρξει επανάσταση επίσης στην γεωργική μας πολιτική με ένα νέο νέο σχέδιο για την γεωργία και με αλληλεγγύη. Η Παγκόσμια Τράπεζα επίσης πρέπει να βοηθήσει στην οικολογική μετάβαση και να, γίνουν και, να υπάρξουν και μέτρα δημοσιονομικά κατά της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Να λοιπόν κάποια σχέδια που καταθέτουμε εμείς σήμερα για την οικολογική μετάβαση. Αυτά περιμένει ο πλανήτης και οι συμπολίτε μας. Ένα σύμφωνο για το μέλλον. Έχετε τρεις μήνες πριν δημοσιευθεί η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει το δικό του ρόλο και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ξαναπεράσει εξετάσει για να αλλάξει επιτέλους το σύστημα και όχι ο πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ. Εύη εκ μέρου των μη εγγεγραμμένων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2005 είναι καλός, αλλά οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί όπως κυκλική οικονομία, η επαναφορά του καθαρού αέρα, αυτά προκαλούν πάρα πολλές αμφιβολίες. Πρώτον, πού θα βρούμε τους οικονομικούς πόρους για να επιτύχουμε την κλιματική αλλαγή και μετάβαση, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι ε, θέλει να επενδύει 260 δις το χρόνο και μετά το ελεγκτικό συνέδριο πριν από λίγο είπε ότι 1150 δις το χρόνο πρέπει να επενδύονται μέχρι το 2030 για να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Άρα δηλαδή ε, κυρία Πρόεδρε φοβάμαι ότι είμαστε πολύ μακριά από το στόχο μας. Είμαστε μπροστά σε μια μοναδική πρόκληση που και εσείς το συγκρίνετε με τον πρώτο άνθρωπο στο ε, φεγγάρι. Πάντως πρέπει να υπάρχουν οικονομικοί πόροι. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει αρκετό θάρρος ούτε για τις πλαστικές ουσίες όλα αυτά που έχουν ληφθεί τα μέτρα δεν φτάνουν. Ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μιλάμε για τα ε, σωστά μέτρα όπως αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί ο κύριος Γιούγκερ. Και ποιος είναι ακριβώ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αντιμετωπιστεί η κλιματική πρόκληση. Τέλος και κλείνω. Αν θέλετε να είσαστε σοβαροί ε, θα πρέπει να ασχοληθείτε κυρίως με την ανάπτυξη γιατί αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Πίπερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την ε, πρόσκληση για πιο φιλόδοξους στόχους. Ε, εάν τελικά επιτύχουμε στην ενεργειακή αλλαγή, τότε η Ευρώπη έχει πάρα πολλές δυνατότητες να επεκτείνει τη βιομηχανία της. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πράγματι προβλέπει μελέτη αντικτύπου για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, να περάσουμε σε νέες πηγές ενέργειας, να δεχόμεθα το φυσικό αέριο ως ε, μεταβατική τεχνολογία. Και αυτά τα χρειαζόμαστε, ε, άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε και δίκτυα για την μεταφορά ε, μέσω αέρα, νερού και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε, πρέπει να έχουμε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες ρεύματο. άρα δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως τις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αλλαγή θα πρέπει να είναι σημαντικό τμήμα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτική γειτονία. Και τέταρτον, η ενεργειακή αλλαγή θα πρέπει να είναι ουδέτερη στην αγορά που σημαίνει ότι ε, αυτά που έχει επιτύχει η βιομηχανία να περάσουν σε κτίρια, ε, να είμαστε ουδέτεροι προ την τεχνολογία, σημαίνει καινοτομίε. Σήμερα ένα αποτελεσματικό αυτοκίνητο diesel είναι πολύ πιο φιλικό προ το περιβάλλον από ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αύριο θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά κυρίε και κύριοι, αυτά τα ε, κρίνει η αγορά και όχι η πράσινη κλιματική και ιδεολογία. Ε, με βάση όλα αυτά χαίρομαι που θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα μισό λεπτό η κυρία Ντάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, τον Ρελέιεν, Αντιπρόεδρε Τίμερμαντ, οι επόμενε χρονιέ είναι το χρονικό περιθώριο που έχουμε στη διάθεσή μα για να προγραμματίσουμε το νέο οικονομικό μοντέλο που θέλουμε να υιοθετήσουμε. Και το ευρωπαϊκό αυτό πράσινο σύμφωνο θα μπορέσει να είναι η επανάσταση που θα βάλει στην πυρήνα του τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μα. Όποιο σχέδιο θέλει πραγματικά να πετύχει σοβαρά αποτελέσματα θα πρέπει να υποστηρίζεται με δεσμευτικού στόχου και μετρήσιμου στόχου, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Πάνε πια οι μέρες που τα κρατημέλη ήθελαν να α, καθυστερήσουν την ανάληψη δράσεως. Για να πετύχουμε αυτά που χρειαζόμαστε μέχρι το 2050 χρειάζεται μείωση σοβαρή του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 και να σκεφτούμε σοβαρούς στόχους για το 2040 μέχρι το 2040. Αυτό δίνει σαφήνεια στα κρατημέλη και στις επιχειρήσεις για το πώς και πότε θέλουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Και καμία, κανένα κλάδο δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από διεθνεί μηχανισμού πολύ απλά για να καθυστερήσει την ανάληψη δρασή. Θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτιλία και την αεροπορία. Οι επιδοτήσει για τα άρρηκτα καύσιμα θα πρέπει να α, σταματήσουν σταδιακά. Χρειάζονται λοιπόν καθαρέ τεχνολογίες για όλου του τομεί και σε όλε τι χώρε. Χρειάζονται καινοτόμου καινοτόμοι τρόποι για να πετύχουμε αυτέ τι επενδύσει. Θα πρέπει να συζητήσουμε πώ θα κινητοποιήσουμε του δημόσιου και δυτικού πόρου προκειμένου να έχουμε τα σωστά έργα και ποιοτικέ θέσει απασχόληση και προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι οι εργαζόμενοι του μέλλοντο για τη μετάβαση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η πράσινη συμφωνία να αποτελέσει το ορόσημο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε δεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί σα για να πετύχουμε και από οικονομική αλλά και από οικολογική άποψη. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, λέει η Πρόεδρο. Δεν έχουμε χρόνο από ό,τι φαίνεται για μπλε κάρτε, μου λένε. Δυστυχώ. Επόμενο ομιλητή για ένα λεπτό, κύριε Καμφάν κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Σήμερα είμαι περήφανο που είμαι Ευρωπαίο. Είμαι περήφανο χάρη σε εσά που είμαι Ευρωπαίο. Γιατί μα παρουσιάσατε σε δέκα ημέρε το πιο ευρύ σχέδιο για την οικολογική μετάβαση για όλη την Ήπειρο. Οι ΙΠΑ αποσύρονται από την Συμφωνία του Παρισιού. Εμεί όμω επιταχύνουμε. Θα είμαστε ω ΡΕΝΙΟΥ στο πλευρό σα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή απόψεων και θέλουμε λοιπόν να αλλάξουν όλα μέχρι αύριο, αλλά δεν είναι αυτό δυνατόν. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στο σχέδιο αυτό, γιατί είναι το μόνο το οποίο θα επιτρέψει και στις επιχειρήσεις ε, και στο περιβάλλον να πετύχουν με την κλιματική ευτεραιότητα μέχρι το 2050. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βλέπουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο μέχρι το 2050, αλλά και ε, απαιτήσει και στόχους το 2030. Θέλουμε λοιπόν να ορίσουμε το, τη μείωση κατά 55% με το 2030 με νομικέ προδιαγραφέ. Είναι σημαντικό λοιπόν να αλλάξετε εσεί του κανόνε των ε, συναλλαγών. Από εδώ και πέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να προσυπογράφει εμπορικέ συμφωνίε αν δεν τηρούνται οι στόχοι του Παρισιού. Είναι ένα νέο τρόπο παγκοσμιοποίηση και άλλο ένα στοιχείο ε, που μα κάνει περήφανο. Και η ομάδα του ΡΙΝΙΟΥ θα είναι στο πλευρό σα, κυρία Πρόεδρε και κυρία Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κυρία Τούσα. Κύριε Βαντελέν, αυτά που προτείνετε πριν από 25 χρόνια θα ήταν υπέροχα. Αλλά δεν είμαστε πριν από 25 χρόνια, είμαστε στο 2019 και είμαστε κολλημένοι στον τοίχο με την καταστροφή μπροστά μα. Χρειαζόμαστε μια νέα πράσινη συμφωνία, η οποία τουλάχιστον 65% να μειώνει τι εκπομπέ ε, αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 τουλάχιστον να σεβαστούμε τη Συμφωνία των Παρισιών. Χρειαζόμαστε μια πράσινη συμφωνία η οποία να γυρνάει την πλάτη στι επιχειρήσει οι οποίε χρησιμοποιούν άνθρακα και να δίνουμε χρηματοδότηση όχι εκεί που καταστρέφεται ο πλανήτης. Μιλάτε για επενδύσεις. Ναι, αλλά δεν είναι 10 δις που χρειαζόμαστε για 10 χρόνια, τα χρειαζόμαστε κάθε χρόνο δεν πάτε αρκετά μακριά, γιατί θεωρείτε ότι η ανάπτυξη είναι η λύση. Δεν πάτε αρκετά μακριά, γιατί πιστεύετε ακόμα ότι πρέπει να βοηθήσουμε τι πολυεθνικέ, τι τράπεζε και το σύστημα το οποίο μα κόλλησε τελικά στον τοίχο. Η πράσινη συμφωνία δεν θα πρέπει να είναι διστακτική, αλλά θα πρέπει να αλλάζει πραγματικά πρότυπο. Η οικονομία πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από τη φύση. Μια πράσινη συμφωνία πρέπει να προσαρμόζει το οικονομικό μα σύστημα και τι συνηθίε μα. Χρειάζονται ισχυρά μέτρα δεσμευτικά με έλεγχο ώστε οι επιχειρήσεις και τα κράτη να σέβονται τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε επίσης ένα κοινωνικό συμβόλαιο και δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. Πρόεδρος, θα κόβω το μικρόφωνο στο μέλλον γιατί πιέζει ο χρόνος. Για δύο λεπτά τώρα ο κύριος Μπορκία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω στην κυρία Φοντελάιν πριν βγει από την αίθουσα ε, δεν ήταν βέβαια κάτι προσωπικό αλλά ήθελα να της πω ότι συμμερίζομαι απλά ένα μικρό κομμάτι όλων αυτών που μας είπε. Ε, για να βελτιωθούμε όμως πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα κρίσιμα θέματα ε, και με πού θα βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό που μοιάζει να είναι το πρόγραμμα Juncker, ε, δηλαδή ισορροπία στον προπολογισμό. Ε, κατά τα άλλα, ε, θέλω να είμαι ο εκπρόσωπο όχι των μεγάλων επενδυτών, θα ήθελα εγώ να είμαι εκπρόσωπο των πολιτών και των επιχειρήσεων που ανησυχούν. Άρα δηλαδή οι φόβοι είναι εκείνοι που μου οδηγούν στο να πω ότι θα έπρεπε όλα αυτά να τα σκεφτούμε πολύ περισσότερο καιρό, να τα έχουμε προγραμματίσει πολύ καλύτερα έτσι ώστε να αποφύγουμε να προβάλλονται τα δαπανηρά απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Ε, να επισημάνουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στην ε, Κίνα, στην παραγωγή χάλιβα. Θα έπρεπε να επιβάλλουμε κάποιους, κάποιες, κάποια πρόστιμα. Αν δεν το κάνουμε θα πνίξουν τη δική μας τη βιομηχανία. Όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα, υπάρχουν προβλήματα τα οποία επιβαρύνουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, έρχονται αντιμέτωπες με την επιθετικότητα του διεθνούς ανταγωνισμού. Μιλάμε επίσης για ε, αγορά, για θέσεις απασχόλησης ε, ε, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες ε, μετεγκαθίσανται και βεβαίω μεταφέρουν και τη ρήπανση. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε το σε δημοσιονομικό πλαίσιο στο πρίσμα, κάτω από το πρίσμα της ε, γεωργίας. Παραδείγματος χάρη θεωρώ ότι πολλές επιχειρήσεις ε, θα κλείσουν αλλά παρόλα αυτά ίσως να έχουν αυτές τις μικρότερες εκπομπές. Εγώ εύχομαι η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ε, δεν μπορείτε να συνεχίσετε γιατί έχετε ε, ξεπεράσει τον χρόνο σας. Και να σας πω και κάτι. Ε, γιατί πάντα εγώ να πρέπει να είμαι εκείνη που να λέω ότι θα πρέπει να κόψουμε τον χρόνο. Έχουμε 20 που έχουν ζητήσει να μιλήσουν στο πλαίσιο τη της διαδικασίας Catch the Eye. γι' αυτό αν συνεχίσουμε έτσι κανείς θα πάρει το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye. Αυτοί που λαμβάνουν τώρα το λόγο να το έχετε κατά νου δευτερόλεπτα θα σας δίνω και ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Ε, κύριε Βόνδρα, ε, κύριε Βόντρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα ακούσει όλα αυτά και δεν κάνει μία ανακοίνωση τύπου. Ε, τι γίνεται με το αποτύπωμα άνθρακα γιατί εδώ πέρα καθόμαστε δύο ώρε. Έχουμε μαζευτεί από όλε τι άκρε τη Ευρώπη και αυξάνεται το α, αποτύπωμα άνθρακα. Ναι, είναι μια ριζοσπαστική α, συμφωνία. Είναι μια πράσινη επανάσταση, αν και το ονομάζουμε συμφωνία. Εμεί είμαστε συντηρητικοί, δεν πιστεύουμε στι επαναστάσει. Ναι, θέλουμε ασφαλώ να συμπεριφερθούμε με υπεύθυνο τρόπο σε ό,τι αφορά τον πλανήτη μα. Θέλουμε να προστατεύσουμε την φύση, είναι καθήκον μα Αλλά το τίμημα δεν μπορεί να είναι να εγκαθαντρήσουμε τέτοιες διαδικασίες ε, που θα επιφέρουν ε, μεγάλο κόστος και θα οδηγήσουν σε άλλη επανάσταση και θα θυσιάσουν ε, το πιο πολύτιμο αγαθό, την συμφιλίωση και την συνεργασία των λαών της Ευρώπης. Δεν πρέπει να είναι μανιφέστο αυτό με πράσινο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, κυρία Μούντικ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. οι συντηρητικοί μπορούν να είναι ήσυχοι. Η πρόταση αυτή δεν έχει να κάνει τίποτε με επανάσταση, δυστυχώς. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές. Πρέπει να μειώσουμε τον άνθρακα. Και όλα αυτά με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Υπάρχουν πολλά καλά, πολλά, πολύ καλά, πολλά καλά στοιχεία στην πρόταση αυτή. Αρκούν όμως για να είμαστε λοιπόν κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, πρέπει να πετύχουμε τους στόχους του 2030. Και οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι φιλόδοξοι. Ήταν, ε, ανακηρύξαμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη σε ό,τι αφορά το κλίμα και μας λένε ότι θα πρέπει οι στόχοι για το 2030 να έχουν μειωθεί οι εκπομπές σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτά που μας λέει η επιστήμη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε μείωση μέχρι το 2030 60%. Ε, δεν φτάνουν αυτά, λοιπόν, που προβλέπονται στο πρόγραμμα, γιατί δεν θα μειωθεί επαρκώ το διοξείδιο του άνθρακα και θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν και η βιομηχανία και η γεωργία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. και τώρα για ένα λεπτό κοράω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ε, θετικά στοιχεία από, με βάση αυτά που ακούσαμε, αλλά εξακολουθώ να έχω πολλές εμφωλίες σχετικά με το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα αυτά που ανακοινώσατε. Έχουμε ε, ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό και όπως αναφέρεται οφείλουμε να παρεμπεδίσουμε ε, το τεράστιο κόστος της μη δράσης. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση, ε, πρέπει να επενδύσουμε τώρα, έχουμε τη φιλοδοξία να, να σώσουμε τον πλανήτη και την αγορά εργασία. αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να επενδύσουμε στην ε, έρευνα, να υπάρχει πρόσβαση στους πόρους, χρειαζόμαστε ένα πιο διαφανή διάλογο με τους πολίτες και πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. Κατά την τελευταία ολομέλεια ανακοινώσαμε την έκτακτη ανάγκη λόγω κλίματος. Αυτή ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια για ευαισθητοποίηση, αλλά πια δεν μπορούμε να περιζόμαστε στα λόγια, χρειαζόμαστε πράξεις και τις χρειαζόμαστε τώρα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαρινέσκου για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Το βρίσκω πάρα πολύ καλό το ότι πλέον έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση. Ελπίζω κατά την επεξεργασία της πρότασης να διαβουλευτήκατε με όλες τις γενικές διευθύνσεις. Δηλαδή η πρόταση αυτή να βασίζεται σε ευρεία συνένεση, σε εφικτές προτάσεις. Καταθέσε τώρα ένα νομοθετικό πρόγραμμα και αυτό το χαιρετίζουμε. Όμως ε, θα ήθελα να παρακαλέσω να εξετάσετε επίσης ε, κατά πόσον ε, όλα αυτά είναι συμβατά μεταξύ τους για να μην ε, προκληθεί σύγκρουση με άλλα νομοθετικά μέτρα. Ελπίζω λοιπόν για όλες τις προτάσεις να υπάρξει μελέτη αντικτύπου τόσο όσον αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής όσο και κάτω από το πρίσμα ε, της ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη. Ελπίζω λοιπόν όλα αυτά να έγιναν μετά από διαβουλεύσεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικέ τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ελπίζω λοιπόν να λάβετε μέτρα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε και τα, τους πόρους του Horizon 2020. Ε, αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη μπορούμε τα κονδύλια αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για την καινοτομία και όχι απαραίτητα για βασική έρευνα. Ε, και να σας παρακαλέσω και κάτι άλλο. Πρέπει να δείτε λιγάκι αυτό το θέμα που αφορά στον πλανήτη, στον κόσμο. Ο κύριος Ερτουκ. Ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ αυτό ε, θα ήθελα να ε, εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον κύριο Τίμερμανς για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε τις τελευταίες εβδομάδες και αγαπητοί συναδελφοί ε, δράτω με τις ευκαιρίες για να καλέσω όλους μας να διεκδικήσουμε αυτή την πράσινη συμφωνία να τη μετατρέψουμε σε μια νέα συμφωνία ένα είδος New Deal της Αμερικής. Τη δεκαετία του 30 κυρίε και κύριοι το New Deal στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα αιτήματα που προήρθαν από την Ευρώπη προκάλεσαν θέσει απασχόληση, οικονομική ανάπτυξη και μια κατεύθυνση προ την κοινωνική ισότητα. Αυτό χρειαζόμαστε για την πράσινη βιομηχανική ανάπτυξη. Οι επενδύσει ε, στι μπαταρίε, ε, ε, στου υδάτινου πόρου, όλα αυτά πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα, πρέπει να υπάρξουν επενδύσει σε σύγχρονε υποδομέ για πράσινη οικονομία τόσο σε μεγάλε πόλει όσο και σε μικρά χωριά. Αυτό είναι λοιπόν ο τρόπο και ο δρόμο δρόμος, με συγχωρείτε, που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κύριος Ντέιβις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς, δεν μπορώ να τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η νέα πράσινη συμφωνία. Ε, πρέπει να σώσουμε τον κόσμο γιατί δηλητηριάζουμε τη Βαλτιδική. Υπεραλλιεύουμε στη Μεσόγειο, καταστρέφουμε προστατευμένε περιοχέ τη. Λέμε ότι είναι προστατευμένε και μετά τι αφήνουμε στην τύχη του. Ε, ψάρια που πετιούνται πίσω στη θάλασσα είναι πεθαμένα, είναι περισσότερα από αυτά που αλλιεύουμε για να τα φάμε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε έτσι. Πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση και να βοηθήσουμε την αποκατάσταση και των ε, αποθεμάτων στη θάλασσα. Η βιωσιμότητα πρέπει να μπει πρώτα απ' όλα και μόνο τότε να κάνουμε διαπραγματεύσει, απαιτώντα και καλή διακυβέρνηση και από του άλλου. Οπότε, κύριε Αντιπρόεδρε, αντιμετωπίζουμε ε, πολλέ μάχε και πολλού αγώνε μπροστά μα. Αυτήν μπορούμε να την κερδίσουμε. Να υποφεληθείτε από αυτή την ευκαιρία, λοιπόν. Έχετε την ευκαιρία και μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση στι θάλασσέ μα και να κάνετε τη διαφορά προ το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. 1,5 λεπτό τώρα ε, ο κύριος Μπούχαϊτ. Α, συγγνώμη. Ένα λεπτό πρώτο, κύριος Νίνιστο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το πήγον του κλίματος είναι μπροστά μας, το ξέρουμε, και η νεολαία στους δρόμους το λέει και μα το υπενθυμίζει και αυτό συζητάμε σήμερα. Και χαίρομαι για την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ήμουνα πρόεδρο περιβάλλοντο και έχω συναντηθεί με διάφορου επιτρόπου και είναι η πρώτη επιτροπή η οποία βάζει τέτοια προτεραιότητα στο θέμα του κλίματο. Αλλά ακόμα δεν είναι αποφασιστική σημασία αυτή η συμφωνία και πρέπει να είναι. Η Πράσινη Συμφωνία και το πρόγραμμά τη είναι υποσχέσει αλλά όχι αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρωτάω λοιπόν είναι διατεθειμένη να φτάσει στο 55% για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων και παραπάνω ακόμα. Είσαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Είσαστε έτοιμοι επίσης να αυξήσετε τους στόχους για την απόδοση ενέργειας. Η ενέργεια βρίσκεται στην καρδιά της μετάβασης που θέλουμε να πετύχουμε. Το 75% μας έρχεται από την ενέργεια των εκπομπών, οπότε η μετάβαση αυτή στην ενέργεια είναι αναγκαία. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για την πράσινη πτυχή. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Μπουχάιτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προέκυψε με τρεις υποσχέσεις. Πρώτον, μείωση των εκπομπών. Δεύτερον, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και τρίτο είναι βελτίωση της ε, ποιότητας ζωής. Το να περιστούν οι εκπομπές, αυτό είναι ένας ε, ευγενής στόχος, αλλά ε, ας μην ξεχνάμε ότι περίπου το 10% των εκπομπών ανά τον κόσμο προκαλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 309 εργοστάσια άνθρακα στην Κίνα. Αυτά ε, θεωρώ ότι είναι ήδη απαρχαιωμένα. Τώρα, κατά πόσον τα μέτρα τη Πράσινη Συμφωνία θα βοηθήσουν, δεν το ξέρουμε. Αυτό που είναι σαφέ αυτή τη στιγμή είναι η περαιτέρω επιβάρυνση ε, και κατακυδεμόνευση των πολιτών μα ε, στην ε, γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Παραδείγματο χάρη, στη δική μου την πατρίδα, με την Audi θα κοπούν πάρα πολλέ θέσει απασχόληση. Άρα, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι και αλλιώ πηγαίνει πηγαίνει προς ύφεση με την Πράσινη Συμφωνία. Εσείς, ε, κυρία Πρόεδρε, ρίχνετε μία τροχοπέδη. Ε, χρειαζόμαστε ελευθερία αντί για επενδύσεις. Χρειαζόμαστε σαφές πλαίσιο, ε, δυνατότητα σχεδιασμού, ασφάλεια, νομική και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σημαίνουν ότι θα πρέπει να τηρούμε την ουδετερότητα της τεχνολογίας προάγοντας μελλοντικά μέτρα. Ε, Επιτροπή, επιτέλους ε, θα πρέπει να αφήσετε ελευθερία στις επιχειρήσεις μας για να μπορούν μόνες τους να αποφασίζουν και εσείς να περιορίσετε τη φαντασία σας. Ο κύριος Ευχιώκη για ένα λεπτό. Αγαπητή κυρία Μαγκίνη ε, και αγαπητή απούσα ε, κυρία Φαντελάιν ελπίζω αυτό να μην είναι μια ένδειξη του τι μας περιμένει, να πιστεύει ότι η ε, πρόεδρος δεν χρειάζεται να ακούει ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο. Θέλω να σας πω ότι κατά 110% στηρίζω την Πράσινη Συμφωνία, αλλά έχω μεγάλες απαιτήσει εσείς προς την απούσα κυρία Βαντελάιν έναντι των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ινδίας. Αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο μας γιατί αν δεν γίνει αυτό αυτή η νέα πράσινη συμφωνία θα είναι άχρηστη, αντιπαραγωγική και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα σχέδια ε, που έχετε εκπονήσει κατ' ουσίαν θα πρέπει να βάζουν τις θέσεις απασχόλησης ως πρώτη προτεραιότητα γιατί δεν θέλουμε όλες οι βιομηχανίες να εγκατασταθούν στην Αφρική, στις ΗΠΑ ή στην Τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό, Μποτένια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κάτι για φιλοδοξία, αλλά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα ε, απογοητεύσετε κάποιου ανθρώπους, όπως για παράδειγμα κάποιου ανθρώπου που ξεκίνησαν να δουλεύουν στα 15 του και πλέον ε, μετά από τόσα χρόνια έχουν ένα σύνταξη 570 ε, ευρώ. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Αυτή ακριβώ ε, οι φόροι είναι για του οποίου διαδηλώνουν οι Ζηλεζούν και όλοι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη. Και μιλάμε λοιπόν για 500, για τόσο πολλά εκατομμύρια εκατομμύρια που ζουν σε καθεστώ φτώχεια. Δεν, ξέρουν να, δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι του. το χειμώνα. Δεν μπορούν να άψουν το φω. Είναι λοιπόν πραγματικά απαράδεκτο να ζητάμε από του ανθρώπου αυτού να πληρώσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα απογοητεύσετε και την Απολύν. Μία φοιτήτρια η οποία κάθε εβδομάδα βγαίνει στον δρόμο και διαδηλώνει κατά των ριζοπλαστικών αυτών μέτρων και βλέπει ότι μιλάτε για επενδύσει, αλλά δεν σταματάτε αυτή την στρατηγική λιτότητα για την ενέργεια δεν σταματάτε το σύστημα ETS για την εμπορία των ρήπων. Πώς μπορείτε να μας τα εξηγήσετε λοιπόν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κ. Σαλαβάνος. Σε περίοδο σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε εμπεριαλιστικά κέντρα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΙΠΑ, Κίνα, Ρωσία, αλλά και σε κολοσσούς της ενέργειας, το Green Deal είναι η απτή απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να δοθεί άφθονο χρήμα στους μεγάλους ομίλους στην κούρσα με τους ανταγωνιστές τους. η ευρωπαϊκή ένωση επιβραβεύει τα μεγάλα συμφέροντα που ρηπαίνουν το περιβάλλον με πράσινα ταμεία και επενδύσεις ύψους τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 ενώ τιμωρεί τις λαϊκές οικογένειες με κάθε έμπνευση πράσινη φορολογία καλλιεργώντα την επικίνδυνη αντίληψη της ατομικής ευθύνης. οι πραγματικές ανησυχίες των λαών για την προστασία του περιβάλλοντος δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα εμπορίου ρήπων με τις εξαγωγές απορριμμάτων με τη λογική ο ρηπαίνων πληρώνει λογικές που ανακυκλώνουν μόνο τα προβλήματα. οι καπιταλιστές και οι ενώσεις τους για το μέγιστο κέρδος εμπορευματοποιούν και καταστρέφουν το περιβάλλον. γι' αυτό επιβαρύνουν το κλίμα. μόνο μια σχεδιασμένη κεντρικά οικονομία χωρί εκμετάλλευση υπεριαλιστικού πολέμου και μονοπόλια μπορεί να ικανοποιήσει τι σύγχρονε κοινωνικέ ανάγκε να εξασφαλίσει τη ζωή και την υγεία του πληθυσμού την προστασία του περιβάλλοντο. For one and a half. Για ένα λεπτό, η κυρία Μόσερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα κατά ε, της κλιματικής αλλαγής πρέπει να ακολουθήσουμε τον Γιούγκερ, τον Αρία Σκανιέτε, τη Συμφωνία των Παρισίων. Αλλά πρέπει να πείσουμε και να απαιτήσουμε όλες τις περιφέρειες ε, του κόσμου να έχουν την ίδια φιλοδοξία όπως έχουμε και εμείς. Εμείς εξάγουμε την χρηστή μας ε, διαχείριση, το know-how μας για να έχουμε έναν ε, πλανήτη που να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Πρέπει να καταπολεμήσουμε λοιπόν την κλιματική αλλαγή και ο καλύτερος τρόπος είναι η υπό την ηγεσία τη Ursula von der Leyen. Αλλά αυτό ο μεγάλο παγκόσμιο στόχο, που είναι στόχος ολονών μα, δεν φτάνει γιατί έχουμε την άρνηση από την άκρα δεξιά και την ιστερία τη άκρα αριστερά. Ο στόχο μα απαιτεί ενότητα, ε, υπευθυνότητα και να μην ξεχάσουμε κανένα στον αγώνα αυτών. Πρέπει συγχρόνω να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, καλύτερε και περισσότερε θέσει απασχάληση, να λάβουμε υπόψη μα όλου του παραγωγικού τομεί και όλου του ε, πολίτε, του ε, ανεξάρτητου επαγγελματίε, του αγρότε, του ψαράδε, τι οικογένειε. Όλου, όλε αυτέ οι οικογένειε επηρεάζονται από την ε, αλλαγή που θέλουμε να πετύχουμε. Και για όλους αυτούς πρέπει να βάλουμε στη διάθεσή μας όλα τα εργαλεία, κοινωνικά, οικονομικά, ε, τα πάντα, νομικά και ε, τις μελέτες αντικτύπου για να μην ξεχάσουμε κανένα. Και ένα μήνυμα προς την νεολαία που είναι το μέλλον του κόσμου. Η καλύτερη σύμμαχή μας ε, στο ΕΛΚΕ είναι ακριβώς η νεολαία υπέρ του πλανήτη και πάντα εμείς ήμασταν πρωταγωνιστές των μεγάλων μεταβάσεων και των μεγάλων αλλαγών. Ευχαριστώ. Η κυρία Φρίτσον, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Τίμερμαντσα, ε, Επιστρέψαμε από τη Μαδρίτη, όπου γίνονται διαπραγματεύσει για το μέλλον μα. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη δεύτερη κλιματικά ήπειρο αυτό σε τοπικό, περιφερειακό και ε, εθνικό επίπεδο, αλλά και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες λοιπόν θέλουμε να αναλάβουμε τον ηγετικό αυτό ρόλο. Η Ευρώπη θα πρέπει να σημειώσει μια μετάβαση οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να έχουμε ίσους όρους. Στην Σουηδία είχαμε μια κυβέρνηση η οποία ε, ψήφισε σχετικά νομοσχέδια και στη Φιλανδία και στην Δανία ψήφισε η κυβέρνηση πολύ φιλοδόξο πρόγραμμα για το κλίμα. Η πράσινη καινοτομία, οι πράσινε θέσει απασχόληση, ε, εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε. Πράσινη ανάπτυξη, αυτή η πράσινη συμφωνία, η οποία θα αποτελέσει το μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μα. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, η κυρία Τσε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή και πολλά υποσχόμενη παρουσίαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαίνεται ότι οι περασμένε γενιέ αγνοούσαν και παραμελούσαν το σχέδιο αυτό. Αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή φαίνεται να προωθεί. Θέλω να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα σχέδια για να πετύχουμε αυτή την ιστορική, το ιστορικό επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Δεν είναι απλό. Είναι έτοιμη η συμφωνία, είναι έτοιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι έτοιμο το Κοινοβούλιο και το Renew Europe. Είναι αλλα Αλλά έχουμε τρία κράτη-μέλη ακόμα που μπλοκάρουν του στόχου τη κλιματική ουδετερότητα ακόμα, συμπεριλαμβανομένη και τη χώρα μου, τη Ουγγαρία. Δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι ότι θα πετύχουμε ένα πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα έχει τι σωστέ προδιαγραφέ. Και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η πραγματική κλιματική δράση δεν θα είναι όμοιρο των πολιτικών συμβιβασμών και θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην υπόσχεση αυτή ενό βιώσιμου μέλλοντο για όλου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκίγκολτ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σήμερα θέλω να σας πω ότι ευχαρίστω είμαι Ευρωπαίος. Είναι μια πολύ καλή ημέρα παράλληλα με την κλιματική διάσκεψη στο Παρίσι. Ε, αυτό είναι καλό ε, και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η προστασία του κλίματος είναι η προϋπόθεση για θέσεις απασχόλησης, για ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και όχι το αντίθετο. Ε, δεν πρέπει να μας ε, φρενάρουν αυτοί που θέλουν μονίμως να παραμείνουν στο παρελθόν. Τώρα έχω αμφιβολίες αν είναι ικανοποιητική η κοινωνική ατζέντα. Πράγματι πρέπει να αλλάξει ε, το θέμα του εμπορίου των εκπομπών. Όμως από την άλλη τα έσοδα από αυτό αυτούς τους φόρους θα πρέπει να επιστραφούν πίσω στους φορολογούμενους κατά κεφαλή, γιατί αλλιώς δεν θα κερδίσουν οι άνθρωποι. Και μια τέτοια ισχυρή κοινωνική διάσταση λείπει στις προτάσεις σας. Κατά τα άλλη, εμείς θα στηρίξουμε τις προτάσεις σας, θέλουμε περισσότερες φιλοδοξίες στην εμπορική, γεωργική, χημική πολιτική, αλλά γενικά είσαστε ε, στον καλό δρόμο και πλέον ας περάσουμε στην πράξη. Για δύο λεπτά ο Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Ζούμε μια στιγμή πράγματι σημαντική και είναι η πρώτη φορά που εδώ στο Σώμα οι οικονομικές και πολιτικές μας ε, επιλογές υπόκεινται στις επιστημονικές και οικολογικές ε, επιλογές. Όμως δεν υπάρχει μόνο μία ε, διάσταση. Υπάρχει η δηλητηρίαση του αέρα και των υδάτων, υπάρχει Υπάρχουν συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών που επίση έχουν μεγάλη σημασία. Και να ξέρουμε ότι όταν σταματάει η βιοπικιλότητα και μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών, είναι κάτι επίση σημαντικό, ίσω και πιο σημαντικό από την εξαφάνιση τη βιοπικιλότητα στα φυτά και τα ζώα. Να ξέρουμε ότι μόνο τα εδάφη μας μπορούν να κάνουν την αλλαγή. Θέλουμε κοινωνίες οι οποίες να προστατεύονται και μόνο τότε μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, και την οικολογική αλλαγή και το επίγονο της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις κοινωνίες και τότε θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε επόμενες γενιές έναν πλούσιο πλανήτη. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν να είμαστε προσεκτικοί από πολλές απόψεις. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις ρυθμίσει, Να μην είναι σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν την μεγαλύτερη δραστηριότητα οικονομική στον πλανήτη μας. Επίσης πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε πίσω από την Πράσινη Συμφωνία να μην κρύβεται η παγίδα της ομοιομορφίας πρακτικών και μεθόδων παραγωγής που θα κατέστρεφαν τις παραδόσεις μας και τις διαιτερότητες των δικών μας ε, περιφερειών που αποτελούν και τον πλούτο της Ένωσης και μπορούν να αντιμετωπίσουν και την ενεργειακή ε, πρόκληση. Έπειτα, προσοχή πώς θα μεταχειριστούμε τα πυρηνικά. Για τα πυρηνικά, για στρατιωτικό και μη στρατιωτικό σκοπό συνδέονται. Είναι το μέλλον μας και είναι αυτό που εγγυάται και την ε, στρατηγική ανεξαρτησία της Γαλλίας. Η συζήτησή μας πρέπει να οδηγήσει να γίνει επιθυμητό αυτό το οποίο είναι και αναγκαίο. Σα εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την πρόκληση. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό, κύριε Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ε, Αντιπρόεδρε Τίμερμαντς, ε, χρειάζονται λοιπόν κατεπηγόντως ε, τα περαιτέρω βήματα για την εκλογική βιδαιότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως σήμερα πιο πολύ είναι συγκεκριμένες λύσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν και θα μπορούσαμε να τις χρηματοδοτήσουμε. Κυρίως θα πρέπει να πετύχουμε λοιπόν την καινοτομία και προτείνεται πραγματικά ένα σχέδιο το οποίο είναι πολύ ε, περιεκτικό, αυτό είναι πολύ θετικό, το οποίο θα προωθήσει και θα εντάξει και την επιχειρηματικότητα και ε, το κλίμα και όλα αυτά. Αυτό που λείπει ωστόσο είναι μια βάση χρηματοδοτική. Συγκεκριμένα σχέδια για τη χρηματοδότηση, τα οποία να βγάζουν νόημα. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα διπλό ρίσκο. Από τη μία, να μην πετύχουμε στην τελική ανάλυση του στόχου σας. Αυτό λοιπόν σίγουρα είναι ο κίνδυνος και επίσης ε, στην πορεία να χάσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τέλος, 10% ούτε καν 10% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προέρχονται από την Ευρώπη. Αυτό ξεχνά το, ξεχνάμε. Ε, θέλετε λοιπόν να είστε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε γεωπολιτικό επίπεδο, άρα να το συμπεριλάβετε αυτό παρακαλώ στη γεωπολιτική σας αποστολή. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Γκιονγκώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και χαίρομαι που βλέπω ότι σε ό,τι αφορά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις η αλλαγή του κλίματος έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ιστορικό το βήμα αυτό και χαίρομαι που συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση για την πρόταση για την Πράσινη Συμφωνία. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η Ευρώπη στη συζήτηση αυτή θα πρέπει να είναι ηγετική φυσιογνωμία σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά φιλόδοξου στόχου, αλλά οι οποίοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, μετρήσιμοι και εφικτοί. Όχι μέχρι το 2050, αλλά πολύ νωρίτερα, κατά πάσα πιθανότητα, μέχρι το τέλος της θετίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξουν και κάποιοι ενδιάμεσοι στόχοι, με τους οποίους θα είναι υπόλογη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους στόχους που θέτει. Και ασφαλώς θα πρέπει να δηλώσουμε ότι έχουμε σπαταλήσει μία δεκαετία και παραπάνω όταν οι παγκόσμιες οικονομικές αγορές είχαν μεγάλη ρευστότητα. Θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν λειτουργικούς στόχους και λειτουργικά προγράμματα βάσει των οποίων θα μπορέσουμε να επενδύσουμε και να προχωρήσουμε στο μέλλον. Και κόπτη η Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ ο κύριος Λίντς για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, μπορούμε να είμαστε περήφανοι, γιατί σήμερα καταθέσαμε ακούσαμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ε, Πράσινη Συμφωνία για το 2050. Οι στόχοι που έχουμε πετύχει ως τώρα όμως δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν. Θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για όλους τους τομείς και για την τεχνολογία και την ηγεσία μας ε, σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ, τα αέρια του θερμοκηπίου, θα πρέπει να υπάρξει όχι μείωση, αλλά να αξιοποιήσουμε και δυνατότητε αποθήκευση. Κανώ ορίζω λοιπόν το γεγονό ότι πέρα από τι άλλε στρατηγικέ ε, έχουμε και μία φιλόδοξη στρατηγική για την διαχείριση ε, των δασών και των αγρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωργία δεν είναι τόσο τμήμα ε, του προβλήματος όσο το τμήμα της λύσης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σωστή διαχείριση αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια ακριβής μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα φυτοπροστατευτικά να μην λαμβάνουμε λαθασμένες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύρια Αντιπρόεδρε, με τους ε, συναδέλφους από τους Σοσιαλδημοκράτε. Ε, σήμερα επανέλθαμε από τη Μαντρίτη όπου τρέχει η Διεθνή Διάσκεψη για το κλιμα COP25. Θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να χαμηλώσει τα μάτια και να βλέπει όχι μόνο το τι κάνουν ε, οι νέοι γιατί διαδηλώνουν και θέλουν ένα πιο καθαρό πλανήτη πλανήτη, να δίδεται μεγαλύτερη σημασία στον ε, πλανήτη μας, αλλά και ο οικονομικός κόσμος ε, χαμηλώνει και αυτό στα μάτια γιατί βλέπει τι γίνεται με αυτή τη νέα συμφωνία. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αποφασιστικότητα του κυρίου Τίμερμανς, ε, ο οποίος αποφάσισε να αγωνιστεί για την κυκλική οικονομία, αγωνίζεται κατά των πλαστικών υλών. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Τώρα, για τα γεγονότα. Δύο πράγματα να πω. Πρώτον, όσον αφορά τους πόρους. Αν θέλουμε μία βιομηχανία με λιγότερη ρήπανση, αν θέλουμε ηλιακούς ε, θερμοσύφωνες και ανακυκλώσιμα ε, υλικά, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές επενδύσεις. Άρα δηλαδή να υπάρχει Συγγνώμη, πρέπει να σας ε, διακόψω. Για ένα λεπτό, κύριος Φέντερλε. Ε, αυτή η πράσινη συμφωνία ε, μπορεί να είναι το ξεκίνημα για μια νέα κατάσταση στην Ευρώπη. Ε, αν τα αντιμετωπίσουμε όλα, όλοι μαζί θα έχουμε νέες επενδύσεις, νέα τεχνολογία και αυτά θα αποτελέσουν την έναρξη μιας νέας εποχής, της πράσινης εποχής. Θα περνάμε από την οικονομία των ρηκτών καυσίμων στην πράσινη οικονομία. Αυτό που λείπει μέχρι τώρα στο έγγραφο είναι η βιοοικονομία η οποία μας προσφέρει τεράστιες δυνατότητες να ξεφύγουμε από τα χημικά, από υλικά των ορυκτών καυσίμων προς υλικά που, είναι πράσινα. Και αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία, θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα βοηθήσει να έχουμε μια νέα έκρηξη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, αυτή λοιπόν η πρόταση, αντί να μειώσει, να συρρυκνώσει, θα αναπτύξει την οικονομία, νέες βιομηχανίες, νέες θέσεις απασχόλησης. Να έχουμε ηγετικό ρόλο, να δείξουμε στον κόσμο ότι μια τέτοια σύγχρονη οικονομία μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό ε, με τις ε, βιολογικές δυνατότητες που μας προσφέρει η φύση. Κυρία Φίλιπς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στις τελευταίες εκλογές είχαμε πολλούς πράσινους ευρωβουλευτές που εκλέχτηκαν και εκατομμύρια διαδηλώνουν για την προστασία του πλανήτη και είναι όλα βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ακολουθεί επιτέλους το δρόμο που χαράξαμε και μιλάει πράσινα. Η δικιά της πράσινη συμφωνία όμως πρέπει επίσης να κάνει το ίδιο. Η πράσινη συμφωνία μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά όχι και νέα. Κύριε Τίμερμαντς, έχετε την ευκαιρία μπροστά σας να αντιμετωπίσετε τις τρεις κρίσεις της Ευρώπης, της ανισότητας, τη δημοκρατική κρίση και την κλιματική κρίση. Χρειάζεται μια πραγματική πράσινη συμφωνία που να αντιμετωπίσει και τις τρεις αυτές προκλήσεις, που να συνδέεται με τον κόσμο, σε αυτό το ταξίδι που θα πρέπει να ακολουθήσει μαζί με τον κόσμο και να αυξήσει τις προδιαγραφές για την ποιότητα της ζωή. Πρέπει να αντιμετωπιστεί λοιπόν η κλιματική αλλαγή και αυτή η πράσινη συμφωνία δεν πρέπει να είναι ένα πρόσχημα. Πρέπει να δώσει αποτελέσματα, πραγματικά αποτελέσματα στου Ευρωπαίου πολίτες. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, Ρόλαντ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μακίνε, οι πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποτύχει, έχουν οδηγήσει σε ψηλές τιμές ενέργειας, ε, περισσότερο από την ε, Αμερική, όπου είναι κατά 8% πιο χαμηλές. Η Ευρώπη λοιπόν πληρώνει τη νύφη. Η οδηγία για τις ανώσιμες πηγές επίσης οδηγεί σε καταστροφές γιατί καταστρέφονται ε, πουλιά τα οποία κυκλοφορούν γύρω από τις ε, ανεμογεννήτριε, οι οποίες επίσης με τη σειρά του κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει τεράστιο λόμπι εδώ στις Βρυξέλλες. Η βιομάσα είναι που, κάτι που δείχνει την υποκρισία και την ηλικιότητα. Έχουμε ηλεκτρισμό επίσης από ξύλα τα οποία εισάγονται από την ε, Αριζόνα. Τελικά Αυτά κοστίζουν 850 εκατομμύρια στους ε, φορολογούμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η πράσινη συμφωνία θα οδηγήσει σε αποβιομηχανοποίηση. Θα καταστρέψει τη φύση και τις οικονομίες της Ευρώπης. Το κρίμα είναι στα χέρια σας. Ευχαριστούμε. Το Μπέ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς οι Σουηδοί Καλωσορίζουμε το Green Deal, αυτή την πράσινη συμφωνία. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρώπη να είναι φιλόδοξη και πιο φιλόδοξη από ό,τι ήταν σε ό,τι αφορά το κλίμα. Αλλά αυτό που θα είναι καθοριστικό είναι τι θα κάνουμε, αν πραγματικά θέλουμε σταδιακά να καταργήσουμε τα ορεικτά καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να δαπανίσουμε πολύ πιο πολύ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρειαζόμαστε επίσης και πυρηνική ενέργεια χωρί διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό θα είναι σημαντικό στοιχείο σε πολλά κράτη-μέλη και γι' αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται για ένα πολύ βασικό στοιχείο αν θέλουμε να πετύχουμε τους ε, φιλόδοξους στόχους μας, γιατί αν θέλουμε η Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, θα πρέπει η κλιματική πολιτική μας να συνοδεύεται από μια ε, ευημερία και ανάπτυξη για να δημιουργήσουμε μια πολιτική η οποία θα υποστηρίζεται και από τους πολίτες στην Ευρώπη. Τότε μόνο αυτό μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Φερνάνδες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για το έργο σας τελευταίες εβδομάδε και συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ανακοίνωση αυτή. Ένα θέμα όμως θέλω να θίξω. Το οικονομικό σχέδιο αυτής, αυτών των νέων στόχων πώς έχει. Φαντάζομαι ότι έχει δει τις προτεραιότητες και τις έχει εκφράσει και ποσοτικά η Επιτροπή. Όμως τι δυνατότητες υπάρχουν για ένα δίκαιο όριο σε σχέση με τις αγωγές που κάνουμε και που προέρχονται από μεγάλες εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα. Τελικά κινδυνεύουν έτσι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές που ήδη κάνει και αυτές που θα κάνει στο μέλλον. Στην ανακοίνωσή σας λέτε ότι βλέπετε ένα κίνδυνο που μπορεί να υλοποιηθεί και ότι εφόσον η υλοποιηθεί, τότε θα φροντίσετε για μέτρα. Μα αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία τώρα, ήδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μίλλερ. Ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, με τις προτάσεις σας θίγετε δύο θέματα που ε, τα έχουν στερνιστεί. Πρώτον, χαίρομαι πάρα πολύ ε, που ανακοινώσετε μια νέα στρατηγική για τα δάση, όμως ε, με προβληματίζει το εσείς δίνετε σημασία μόνο στην αναδάσωση. Η αναδάσωση είναι μια έννοια που δεν έχει οριστεί ακριβώς και πρέπει να συζητήσουμε επ' αυτής. Εκτός αυτού, η νέα δασική στρατηγική θα πρέπει να προβάλλει ε, τον πολυλειτουργικό ρόλο των ε, δασών. Δεύτερον, η πολιτική από το χωράφι στο πιάτο. Εγώ περίμενα μια διαφορετική στρατηγική. Τώρα όμως βλέπω μόνο επιπρόσθετες υποχρεώσεις για τους γεωργούς. Και η στρατηγική δεν ξεπερνάει το χωράφι, δεν ξεπερνάει την αγροτική καλλιέργεια. Λείπουν άλλες πολιτικές για τους γεωργούς ε, και επίση και λείπουν και άλλα βήματα της αλυσίδας εφοδιασμού η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο θέμα παραγωγής αλλά είναι και θέμα μεταποίησης εμπορίου, εισαγωγών ε, και ενημέρωσης των καταναλωτών. Ε, το δρόμο μέχρι το πιάτο κύριε Πρόεδρε ε, πρέπει ακόμα να τον συμπληρώσετε. Ο κύριος Κόφ για ένα λεπτό. Ε, κύριε Βαντελάν, κύριε Τίμερμαν, σήμερα ε, κάνετε ένα σημαντικό βήμα στο να παρουσιάσετε το, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Χαιρόμαστε γι' αυτό, το περιμέναμε αρκετό καιρό. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι η κλιματική πράξη ε, κοστίζει πολύ, απειλεί την ελευθερία μας, ότι προχωράει αργά. Πρέπει να ξεπεράσετε όλα αυτά, να είστε πάνω από όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί κανείς να βάλει τιμή σε ένα πλανήτη που είναι βλαβερός για τα παιδιά μας. Στην Ιρλανδία 140.000 παιδιά ε, ζουν σε σπίτια απαράδεκτα, με μούχλα, με διαρροές. Εμείς θέλουμε μια νέα συμφωνία στην Ευρώπη που να προσφέρει ζεστά σπίτια, να αντιμετωπίσει τη φτώχεια, να σπάσει τον φαύλο κύκλο της φτώχειας. Στην Ευρώπη 500.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν από ε, κακή ατμόσφαιρα, κακό αέρα. Να προάγεται λοιπόν τις ανάσχημε πηγέ ενέργειας, ε, να σώσει τον ο Επίτροπος Μεταφορών ε, αναφέρθηκε ε, στα ε, αεροσκάφη. Γιατί όμως αυτά να έχουν προτεραιότητα έναντι των τρένων και άλλων μέσων μεταφοράς. Επόμενη είναι η κυρία Νταματό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, Ανακοινώστεται αυτό το η νέα πράσινη συμφωνία ως ένα είδος κατεπήγων, αλλά εξαφανίστηκε η Πρόεδρος. Αν ε, ε, αυτό είναι ο σεβασμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, την, για τον μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμό, λυπάμαι πάρα πολύ. Ανησυχούμε, ανησυχούμε πάρα πολύ. Αυτά είναι μόνο υποσχέσεις. Κύριε Τίμερμαν, η δική σας επιτροπή δεν μπορεί να λέει ότι θέλει να ζήσει σε ένα υγιές περιβάλλον, να τρώει ε, υγιή τρόφιμα, ε, ότι δεν απειλείται. Το δικό σας το πρόγραμμα, ε, λυπάμαι θα το πω, δεν αρκεί γιατί την πραγματική επανάσταση πρέπει να την κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορεί να είναι επανάσταση αν δεν συνεχίσουμε την ανάπτυξη. Έχω κατά νου μακροοικονομικούς κανόνες που θα βοηθήσουν στην πράσινη ανάπτυξη, που θα βοηθήσουν στο να φύγουμε από τον άνθρακα, να προάγουμε το αέριο. Ε, το Transition Fund ε, δεν μπορεί ε, να είναι απλά κάτι για να μας καθησυχάσει. Πρέπει να έχουμε μέτρα έκτακτης ανάγκης. Διακόπτεται η ομιλία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαντς. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν προσυπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού. Η πράσινη συμφωνία λοιπόν αυτή είναι κάτι το οποίο χαίρει γενική υποστήριξη και όλοι οι κλιματικοί στόχοι άλλωστε. Το θέμα δεν είναι μόνο το κλίμα, το θέμα είναι η καθαρή ατμόσφαιρα, οι καθαρέ ε, θάλασσε και οι καθαροί ωκεανοί. Αυτή η πράσινη συμφωνία ουσιαστικά θέλουμε να καταδείξει ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και ότι η οικονομία μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόληση. Και να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να έχουμε ένα, μια χρυσή τομή και αυτή να ακολουθήσουμε. Καταρχάς, να σκεφτούμε τι γίνεται μέχρι το 2030. Στη συνέχεια, χρειάζεται και μια ανάλυση για το τι συνέπειες θα έχουν όλα αυτά. Και να μην ξεχνάμε τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ένα ειδικό πρόγραμμα. Και το έχω υπόψη μου. Και διακοπτή πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ροντρίγκης Ραμός. Νομίζω ότι είναι, εγώ είμαι ο κύριος Νίκα. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε πάλι. Ο κύριος Νίκα και μετά η κυρία Ροντρίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, σας συγχαίρω για την πρότασή σας σήμερα. Πρόκειται για ένα πολύ ε, ευρύ πακέτο, το οποίο είναι πολύ ελπιδοφόρο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών. Και εδώ ορίζεται κάτι σημαντικό, ότι όλοι οι πολίτες και όλες οι περιφέρειες θα πρέπει να υποστηριχθούν. Κανείς δεν μπορεί να μην ξεκρέμαστος. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω να κοιτάξουμε κάποια από τα δικαιώματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία, το κόστος για την επίτευξη των στόχων μέχρι το 2030 είναι 4% του ΑΕΠ. για να πετύχουμε δηλαδή τους στόχους. 8 δις λοιπόν ένα έτος. Μιλάμε για τεράστιο ποσό. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν και τις περιοχές ε, που απασχολούνταν στον Ανθρακά γιατί μιλάμε για 200.000 οικογένειες. Χρειάζεται παράλληλα και ε, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Θα θέλαμε λοιπόν να μας βοηθήσετε προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας το 2030. Τώρα κυρία Ροντρίκης Ραμός λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη εμφάνιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να παρουσιάσει την Πράσινη Συμφωνία είναι ένα σύμβολο για τις προτεραιότητές της και για την πολιτική της αποφασιστικότητα και η πολιτική μου ομάδα την ευχαριστεί γι' αυτό. Χρειάζονται αυτά τα μέτρα, χρειάζονται φιλόδοξα μέτρα. Ε, νόμος για το κλίμα, ενίσχυση της φιλοθεξίας μας για την κλιματική ουδετερότητα του 2050, προστασία των συνόρων, αγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που να είναι καινοτόμα και να μην ρηπαίνει, ε, βιοπικιλότητα, ε, γεωργία. Πράγματι, Πρόκειται για μεγάλους στόχους και για μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτή η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια νέα ε, στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Να είμαστε στην πρώτη γραμμή υπέρ της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της γνώσης, που να είναι πράσινο όμως. Νέες ευκαιρίες επίσης για τις επιχειρήσεις μας. Όλα αυτά σε μια μετάβαση που πρέπει να είναι δίκαια κοινωνική, κοινωνικά και να μην ξεχνάει κανέναν. Σε μια τέτοια στρατηγική δίνουμε τη στήριξή μας κι εμείς. Ευχαριστούμε η κυρία Καστίγιο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Τίμερμαντς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η μάχη κατά της έρμανσης του πλανήτη δεν μπορεί να περιμένει, αλλά ούτε μπορεί και να καταστρέφει. Από αυτή την πλευρά λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε μια βιομηχανική ευρωπαϊκή στρατηγική που να είναι σε θέση να αναπτύξει τεχνολογίες με αποφασιστικό τρόπο να μειώνονται εκπομπές αλλά συγχρόνως να κερδίζει σε ανταγωνιστικότητα παγκοσμίω. Και αυτό απαιτεί να τονίσουμε την καινοτομία με τέτοιο τρόπο που να μπαίνει επίσης ώρες όπως και οι στόχοι της μείωσης των εκπομπών και να εκφράζεται με συγκεκριμένες αποφάσεις όπως μεγάλες προσπάθειες υπέρ της χρηματοδότησης της τεχνολογικής καινοτομίας. Και αυτό είναι το πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας. Σίγουρα στη Μαδρίτη μπορούν να αποφασιστούν πολλά από τις κυβερνήσεις. Εδώ όμως πρέπει να αποφασίσουμε για τον προϋπολογισμό για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. Η Πράσινη Συμφωνία είναι φιλόδοξη. Όλοι συμφωνούμε με την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς να καταστρέφουμε και χωρίς να ξεγελάμε και να ξεγελιόμαστε. Ευχαριστούμε κυρία Μάρκες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για τον αντιπρόεδρο Τίμερμαντς. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να είναι εξαιρετικά φιλοδόξη. Θα πρέπει να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη με δίκαιο τρόπο και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι σωστό για την Ευρώπη τα επόμενα δεκαετία. Αλλά αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με αξιόπιστο τρόπο μόνο αν χρηματοδοτήσουμε με κινητοποιώντα του οικονομικού μα πόρου. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι απαραίτητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Εξετάζουμε το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και η πρόταση την οποία θα συζητήσει αυτό το Συμβούλιο είναι πραγματικά κάτι παραδεκτό. Γιατί είναι εντελώ αντίθετη με τα πολιτικά σχόλια τα οποία εξήγηλαν οι πολιτικοί ηγέτες. Αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε στη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προπολογισμό και αυτή η μετάβαση θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το υποστηρίζουν όλοι. Και όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση και όλοι θα πρέπει να πιστεύουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο κ. Χάιτουμα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι θα πρέπει να λάβουμε δράση κατά τη αλλαγή του κλίματο. Η κατάσταση, οι καιρικέ συνθήκε είναι όλο και πιο ακραίε. Δεν μπορούμε όμω αυτά να μείνουν σε, στα χέρια μιας χώρας ή ενός κλάδου. Θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα και να ακολουθήσει ο υπόλοιπο κόσμος. Μαζί με τους ανθρώπους λοιπόν και με τις επιχειρήσεις θα πρέπει να τα πετύχουμε αυτά. Αλλά μόνο αν καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις αυτές από κοινού. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη από όλου. Δεν έχει νόημα αν δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τους λογαριασμού τους, να μιλάμε για οικονομία και να την ξαναβουτήξουμε στην ύφεση. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν, να περάσουμε από τον πράσινο ιδεαλισμό ε, στην κοινή λογική. Γιατί δεν ζούμε σε μια πραγματικότητα στα χαρτιά. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη αποτελεσματικότητα. Όπω για παράδειγμα το σύστημα εμπορία ρήπων. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην καινοτομία. Γιατί εδώ έχουμε προβλήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, κλίμακα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είτε μα αρέσει είτε όχι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ακολουθήσουμε τι προτιμήσει μα και να αποκλείουμε διάφορε τεχνολογίε όπω την πυρηνική ενέργεια ή η αποθήκευση του άνθρακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πούσο, για έγινε λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε, η αλλαγή κλίματος είναι η πιο μεγάλη και πιεστική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και έχει αντικτύπωση όλο τον κόσμο και επίσης ε, αλλάζουν τα πράγματα γρήγορα. Είμαι αισιόδοξο ότι θα ανταπεξέλθετε στο ύψο των περιστάσεων και ω πρόεδρο τη ΣΥΤΡΕ θέλουμε να πετύχουμε μια συνεκτική πολιτική για την βιομηχανία με μια δίκαιη μετάβαση και να φροντίσουμε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τι προσπάθειέ μα για την ενεργειακή αποβατικότητα, να επιταχύνουμε τι καθαρέ τεχνολογίε, να βελτιώσουμε τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των περιφερειών και να ενοποιήσουμε περαιτέρω την ε, ενιαία αγορά για την ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν στην αγώνα μας αυτόν να κινηθούμε προς την ε, ψηφιοποίηση, την καινοτομία στην, και ε, το κλίμα, να αυξήσουμε τον αριθμό των θέσεων απασχόληση και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί για να υπάρχει ανάπτυξη. Κυρία Φαμπρέμπτη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε οι επιστήμονες έχουν κάνει εδώ και πολύ καιρό τη δουλειά τους και μας έχουν καταδείξει πόσο κατεπήγονται το θέμα αυτό. Και τώρα λοιπόν επιτέλους έχουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για μας αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα μόνο για το κλίμα, μόνο για την αλλαγή του κλίματος. Είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό έργο, όχι μόνο για τα επόμενα χρόνια, αλλά για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό το έργο λοιπόν ουσιαστικά περιλαμβάνει τη δυνατότητα, το δυναμικό να προχωρήσουν προς το εμπρός όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Το δικαίωμα για την καθαρή ατμόσφαιρα, για παράδειγμα, σε όλες τις πόλεις. Όλες αυτές τις θέσεις απασχόλησης, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν για να μπορέσει ο κόσμος να προετοιμαστεί για μια νέα θέση. Να έχουμε υπόψη μας ότι θα μειωθούν οι λογαριασμοί που πληρώνουμε για ηλεκτρικό, γιατί επενδύουμε σε νέα κτίρια. Και αυτό θα πρέπει να το δώσουμε ως μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο και αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό στοιχείο σε αυτή τη νέα πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χλάβατσεκ. Ένα λεπτό. Κύριε... Κύριε Αντιπρόεδρε, η νέα σας πρόταση βασίζεται σε οικονομικά εργαλεία και δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι όλοι θα το διαπιστώσουν. Ε, θέλετε οι πολίτες να σας στηρίξουν, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο αν είσαστε ειλικρινείς όχι μόνο να λέτε αυτά που θα θέλατε, αλλά και για τις επιπτώσεις, να μιλήσετε και για τις επιπτώσεις. Γι' αυτό θέλω να ακούσω από εσάς ότι όλα αυτά που μας είπατε ε, θα τα πλαισιώσετε με μελέτες ε, κοινωνικών και οικονομικών ε, επιπτώσεων. Γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές στην ίδια θέση. Εμείς έχουμε πολλές περιοχές με χαλιβουργία, ανθρακοριχεία, αυτοκινητοβιομηχανίες και αυτοί ενδεχομένως να μην κερδίσουν. Γι' αυτό λοιπόν λοιπόν ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η Ευρωπαϊκή Συνοχή. Καλά όλα αυτά στα χαρτιά, αλλά το θέμα που τίθεται είναι πώς θα επιτύχουμε τους στόχους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ανοιχτοί και στην πυρηνική ενέργεια που δεν ε, ρηπαίνει με εκπομπές. Ε, σας ευχαριστώ πολύ ε, που σέβεστε το χρόνο. Ε, πρέπει να τελειώσουμε το αργότερο μέχρι τις 4 και 10, άρα δηλαδή δεν θα έχουμε διαδικασία Catch the Eye. Λυπάμαι, δεν είναι δική μου απόφαση, απλά ε, δεν έχουμε άλλη λύση. Η κυρία ε, Τότ. Αξιότιμε Αντιπρόεδρε, ε, χαίρομαι πάρα πολύ και το εκτιμώ που καταθέσατε την πρώτη πράσινη συμφωνία γιατί είναι η πρώτη συμφωνία για την προστασία του πλανήτη τα κοινοβούλια προσπαθούν να βρουν κάποιες λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό και εμείς ε, ε, θέλουμε και χαιρόμαστε που υπήρξε αυτή η κλιματική έκτακτη ανάγκη. Αλλά για να πετύχουμε τους στόχους πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο θα ικανοποιεί τους πολίτες, ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα μετακυλεί το κόστος στους καταναλωτές. Οι τιμές ενέργειας και τροφίμων δεν πρέπει να αυξηθούν, άρα ε, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που να είναι αποτελεσματική από το πρίσμα του κόστους και να είναι και ουδέτερη ως προς τις ενεργειακές συνέπειες. Ε, δεν αρκεί να έχουμε μια φιλόδοξη πράσινη συμφωνία. Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες των κρατών μελών, ε, την προστασία του καταναλωτή αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ντεκάστρο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Φραντς, ε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια δύσκολη κατάσταση εμφανίζεται με ε, κλιματικές καταστροφές που πλήττουν τους πελίτες μας. Ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Σήμερα ε, αυτά που παρουσιάστηκαν αναμφίβολα είναι μια πολύ φιλόδοξη συνέχεια. Υπάρχει καταρχήν, ε, θα πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή των ε, γεωργών αν θέλουμε να αμβλύνουμε τις ε, κλιματικές επιπτώσεις γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Πρέπει να κατευθύνουμε τους γεωργούς, να τους δώσουμε κίνητρα για να κάνουν άλλο ένα άλμα στην ποιότητα, να προσφέρουν υπηρεσίες που θα βοηθήσουν το σύνολο του πλανήτη. Αγαπητέ Φράντσε, η πρόταση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής πάνω στην οποία δουλεύουμε. Θα πρέπει να έχει μια στρατηγική που να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση, την επανεθνικοποίηση παρεμβάσεων. Αγαπητέ Φραντς, να έχουμε μια γεωργική πολιτική που να είναι πιο κοινή, πιο ισχυρή, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι το κλειδί για το μέλλον και την ενεργειακή αλλαγή. Ο κύριος Κέλλη τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή που ήρθε εδώ δέκα μόλις μέρες αφού όταν έλαβε τα καθήκοντά της. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν και θα συνεργαστώ μαζί της για να πετύχουμε τους στόχους που μας ανέφερε. Η Πρόεδρος υποσχέθηκε ότι δεν θα ξεχάσουμε κανέναν και ο μηχανισμός που πρότεινε είναι ευρύτερος από ό,τι περιμέναμε και πολύ χαίρομαι γι' αυτό ιδιαίτερα για περιοχές που έχουν άνθρακα όπως είναι τα Midlands και άλλες. Όντως, αν δεν ξεχάσουμε κανέναν θα πετύχουμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τέλος, η χώρα μου μέχρι τώρα είχε μείνει πίσω, αλλά και εγώ και εσείς ε, αντιπρόεδρε και άλλοι συνάδελφοι θα φροντίσουμε να τα καταφέρουμε και να βρισκόμαστε και εμείς στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστούμε. Σαν για ένα λεπτό η κυρία Γιονγκέριους τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η αλλαγή για να φτάσουμε σε μια βιώσιμη κοινωνία θα βοηθήσει και θα γίνει πραγματικότητα αν πράγματι δεν ξεχάσουμε κανένα. Όμω κάποιε κυβερνήσει φοβάμαι ότι δεν θέλουν το ίδιο γιατί αυτή τη στιγμή μπλοκάρουν νομοθεσία στο Συμβούλιο για ε, καθαρή ατμόσφαιρα και καθαρό περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν όλοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας την βιωσιμότητα και για το κλίμα αλλά και για την κοινωνία και να μικρύνει το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση για την φτώχεια αυτή σε σχέση με το περιβάλλον. Υπάρχουν ε, οι άνθρωποι επίση που δουλεύουν στη βιομηχανία. Χρειάζονται θέσει απασχόληση και για αυτού του ανθρώπου που θα ψάχνουν δουλειά στη συνέχεια. Η σημερινή ανακοίνωση πρέπει να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων μας ώστε η πυρός μας πράγματι το 2050 να γίνει ουδέτερη κλιματικά. Φραντς, όσον μας αφορά είσαι ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Η κυρία Φερκίνεν, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αυτή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τον, τρόπο, τον σωστό τρόπο για να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητά μέχρι το 2050 και χαίρομαι ιδιαίτερως που οι διάφοροι τομεί της κοινωνίας έχουν λεφτεί υπόψη σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, τη βιοπικιλότητα, τη βιώσιμη, τις βιώσιμες μεταφορές, τη σχετική νομοθεσία, την εμπορική πολιτική. Είναι σαφέ ότι αν θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι κλιματικά, θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπο που λειτουργεί η οικονομία μα και η κοινωνία επίση θα πρέπει να προσαρμοστεί. Να ενισχύσουμε επίση την καινοτομία στην ε, Ευρώπη, προκειμένου να είμαστε και στο μέλλον ανταγωνιστικοί. Κάποια στοιχεία θα πρέπει να τα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Για παράδειγμα, τους δασμούς, το σύστημα εμπορίας ρήπων. Λοιπόν, χρειαζόμαστε πραγματικά ε, λιγότερες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κυρία Φραν Τίμερμαν, ναι, η αλλαγή του κλίματο αποτελεί μία από τι πιο μεγάλε προ... προκλήσει τι οποίε αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μπορεί να είναι η σωστή απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Συνοχή αποτελεί ένα πιο βασικά επενδυτικά εργαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη τώρα εστιάζεται στα κλιματικά μέτρα. Στο μέλλον αυτό θα πρέπει να είναι πιο έντονο και γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να αντιμορφώσουμε το Μελλοντικό Ταμείο Συνοχή στην παρούσα φάση. Χρειαζόμαστε όμω και πιο έντονη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, τα οποία προ το παρόν είναι πολύ διστακτικά. Θα πρέπει να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να έχει σωστή χρηματοδότηση. Αυτό τι σημαίνει. Δεν μπορούμε να έχουμε λιγότερου πόρου. Αντιθέτω, χρειαζόμαστε φρέσκο χρήμα προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία να έχουν σωστή υποστήριξη σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Χρειαζόμαστε όλου του εταίρου, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, αλλά και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριο Αμάρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η φιλόδοξη συμφωνία η οποία παρουσιάζεται σήμερα χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η πράσινη συμφωνία να οδηγήσει σε ανάπτυξη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε νέε προκλήσει και ότι έχουμε νέε μεθόδου και νέε τεχνολογικέ, οικονομικέ ε, λύσεις και χρειάζονται καινούργιοι πόροι. Το πρόγραμμα από το χωράφι στο πιάτο είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει οι αγρότες να υπάρχουν. Να υπάρχουν τα αγροκτήματα αυτά, αν θέλουμε να έχουμε κάτι να βάλουμε και στο πιάτο μας δηλαδή. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν ο κόσμος να σταματήσει να φεύγει από την Ήπεθρο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο γιατί αδειάζει η πέτρος. Αδειάζουν τα χωράφια και πώς θα έχουμε κάτι να βάλουμε στο πιάτο μας. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει αυτή η αλλαγή και αυτή, το τμήμα της αλλαγής θα πρέπει να είναι και αυτό να ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Αμάρο. Vicepresidente Timmer ο Αντιπρόεδρος κύριος Τίμερμαν Κύριε Τίμερμαν, εσείς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τη συζήτηση ε, και πραγματικά ε, χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι αυτό το Κοινοβούλιο εξέφρασε ευρύτατη συνένεση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτό αποτελεί μια θαυμάσια αρχή ε, σε αυτό που θα είναι ένας ακαθόδη δρόμος γιατί χρειαζόμαστε και οι δύο θεσμοί να εστιάσουν την προσοχή τους σε όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η Πράσινη Συμφωνία. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω το εξής. Ε, θα ήθελα να ε, συγχαρώ την Γκρέτα Τούμπερκ, την οποία το περιοδικό Time ε, την όρισε πρόσωπο της χρονιάς. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα. Τα παιδιά μας μας δείχνουν τον δρόμο. Και ως γονιός πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να βλέπεις τα παιδιά σου να δείχνουν τον δρόμο. Αλλά δεν είναι αυτός ο μόνο λόγος που πιστεύω γιατί πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Το πιστεύω γιατί τα γεγονότα μας λένε ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε κατά πρόσωπο. Και αν λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι, αν είναι κανείς σε υπεύθυνη θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν είναι πολίτης, αν είναι γονιός, δεν έχει κανείς την πολυτέλεια να αγνοεί τα γεγονότα. Για δέστε λιγάκι τι γίνεται στην Γρυλανδία, τι γίνεται γενικά με το κλίμα, με την απερίπμωση, με τον κυκλοθυμικό καιρό. Οι υποφέρουν ε, λόγω αυτού του καιρού. Για δέστε λιγάκι τι γίνεται με τη βιοπικιλότητα τώρα που μιλάμε. Δεν έχουμε λοιπόν την πολυτέλεια όλα αυτά να τα αγνοούμε πια. Και υπάρχει και κάτι άλλο που διαδραματίζεται. Βρισκόμαστε στο μέσο της τέταρτης ε, βιομηχανικής επανάστασης, η οποία θα αλλάξει την οικονομία μας, τη βιομηχανία μας, είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε δραστηριοποιηθούμε είτε όχι. Άρα δηλαδή το ερώτημα που καλούμεθα σήμερα επί του οποίου να τοποθετηθούμε ως Ευρωπαίοι είναι θα μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε, να ελέγξουμε αυτές τις αλλαγές ή θα τα αφήσουμε απλά να ε, εξελίσσονται, άλλοι να τα ελέγξουν και εμείς απλά να είμαστε υποκείμενα που θα δέχονται τις αποφάσεις άλλων. Αυτό είναι το θεμελιώδης ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Και η Πράσινη Συμφωνία δεν είναι ένα σχέδιο, είναι χάρτης πορείας. Σας τίνουμε χέρι βοηθεία και συνεργασία σε εσά, σε όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε είναι βιομηχανίες, είτε ΜΚΟ, είτε συνδικάτα, πολίτες, πόλεις, περιφέρειες. Όλοι να γίνουμε, να συμμετάσχουμε στη συζήτηση για το πώς θα οργανωθούμε ως κοινωνία με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να φαίνονται οι αξίες που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε, γιατί η μητέρα γη κουράστηκε, βαρέθηκε αυτή τη και ξέρετε, η μητέρα γη ήταν εκείνη η οποία τα κατάφερε να επιβιώσει χιλιετίες με όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα. Ε, θα μπορέσει να τα καταφέρει και άλλες επόμενες χιλιετίες ε, και χωρίς ε, ανθρώπινα όντα. Γι' αυτό λοιπόν να συνεχίσουμε την ύπαρξή μας σε ισορροπία με τη μητέρα γη. Και αυτή είναι η ευθύνη που φέρουμε και έχουμε αναλάβει έναντι των παιδιών μας. Να πω και κάτι γιατί αναφέρθηκε επανειλημμένα ότι είναι δαπανηρό. Πράγματι, είναι όλο αυτό δαπανηρό. Για σκεφτείτε όμως πόσο θα κοστίσει το να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Επίσης αναφέρθηκε ότι πρέπει να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν κάθε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνοδεύεται από μελέτη αντικτύπου. Θα είναι αυτό καθοριστικό στοιχείο των αναλύσεών μας. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνουμε με ταχύτητα και κατανοητό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, για να ορίσουμε ακριβώς, ποια θα είναι η μείωση ή πρέπει να είναι μέχρι το 2030 από το 50 μέχρι το 55% θέλουμε να έχουμε μελέτη αντικτύπου αλλά θέλουμε να είμαστε και έτοιμοι στις αρχές του ε, καλοκαιριού του επόμενου έτους έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη με κλιματική νομοθεσία να την παρουσιάσει στην COP26 στη Γλασκόβη να καταδείξουμε τον δρόμο ε, είχα πάει στη Μαδρίτη, θα ξαναπάω αύριο εκεί να τους παρουσιάσω την Πράσινη Συμφωνία και έχω ένα μήνυμα να μεταφέρω. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή ηγεσία και επίσης και εξή μήνυμα. Μερικοί δεν είναι σίγουροι τι πρέπει να κάνουν. Αλλά αν η Ευρώπη καθοδηγεί, τότε θα ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν. Πολλοί λένε ότι η κλιματική ουδετερότητα είναι μια πολύ καλή ιδέα. Οι Κινέζοι λένε θα υπάρχει συλλογική ηγεσία επ' αυτού. Ναι, πρέπει να υπάρχει, γιατί αν προχωρήσουμε μαζί, η ε, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ πιο αισθητά. Και σε τελική ανάλυση αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πει στα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο να κάνουν το σωστό. Αν λοιπόν αρχίσουμε ε, καταγράφοντας ε, ή προσπαθώντας να κατοχυρώσουμε στο, με νόμους ότι μέχρι το 2050 θα είμαστε ε, εκείνοι που θα καθοδηγούν, τότε νομίζω μπορούμε και να φτιάξουμε και το χάρτη που μας οδηγεί οδηγεί σε αυτό το στόχο και θα μιλήσουμε για τα μέτρα. Αν θα είναι για τις εκπομπές, για τη φορολογία ή αν θέλετε οποιοδήποτε άλλο μέτρο έτσι ώστε η βιομηχανία μας να γίνει κυκλική, να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης σε αυτή τη νέα οικονομία. Και να προσθέσω και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι εκείνοι που είναι οι πλέον ευάλωτοι από την κλιματική αλλαγή. Εκείνοι που αντιμετωπίζουν τον τον τους και ως πιο ευάλωτοι στις αντιδράσεις στην κλιματική αλλαγή. Και είναι αυτοί που αρχίζουν να ανθίστανται στην Πράσινη Συμφωνία γιατί αισθάνονται ότι είναι τρωτοί και τελικά ε, θέλουν να σταματήσουν την Πράσινη Συμφωνία. Μα αυτοί θα είναι τα πρώτα από το να μην κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό πραγματικά είναι θεμελιώδες. Αν τελικά δεν έχουμε μια κοινωνική πράσινη συμφωνία, τότε η πράσινη συμφωνία δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Αν δεν υπάρξει πράσινη συμφωνία με τις πλέον ευάλωτες περιοχές Ευρώπης, αν και άλλα, αν δεν υπάρξει αλληλεγγύη από άλλα μέρη της Ευρώπης δεν θα γίνει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε αλληλεγγύη με ευάλωτους πολίτες και ευάλωτες περιοχές για να διασφαλίσουμε ότι η πράσινη συμφωνία θα μπορεί να εφαρμοστεί για όλους τους πολίτες μας και Τελειώνοντας, ο κύριος Λάγκε αναφέρθηκε στον άνθρωπο στο φεγγάρι, γι' αυτό και εγώ μου ήρθε στο μυαλό αυτά που είπε ο JFK, ο Kennedy για τον άνθρωπο στο φεγγάρι. Είχε πει λοιπόν τότε, επιλέξαμε να πάμε, εκείνο και πει στο φεγγάρι, εμείς επιλέξαμε για την κλιματική αλλαγή το 2000 μέχρι το 2050. Όχι διότι τα πράγματα είναι εύκολα, αλλά γιατί είναι δύσκολα, σκληρά, διότι αυτός ο στόχος θα βοηθήσει έτσι ώστε να οργανώσουμε, να καταμετρήσουμε τις ενέργειές μας και τις δεξιότητές μας. Αυτή είναι μια πρόκληση που δεχόμεθα, που δεν θέλουμε να αναβληθεί, μια πρόκληση που προτιθέμεθα να την κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμεί, ε, λέει ο ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμαν. Ε, ευχαριστώ όλους όσοι παρενέβησαν. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία θα γίνει κατά την πρώτη ολομέλεια του Ιανουαρίου. Ε, τα πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στην επόμενη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.